υπάρχουν τροποποιήσεις τη ημερησία διατάξεω, σχόλια κτλ. Όχι, επομένως θεωρείται εγκεκριμένη η ημερησία διάταξη ω έχει και χωρίς καμία τροποποίηση. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει... Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός από εστονικά και μαλτέζικα. Σήμερα εργαζόμαστε για πρώτη φορά με το e-meeting, ηλεκτρονική συνεδρίαση tool. Είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο που αποφασίσαμε πρόσφατα εκείνοι οι συνάδελφοι που χωρίς έγγραφα και έντυπα θέλουν να εργαστούν μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά. Έχετε και εδώ διαφάνεια σχετικά οι συνάδελφοι από τη διοίκηση που είναι αρμόδιοι γι' αυτό λειτουργεί ανεξάρτητα από την πλατφόρμα. Είναι στο διαδίκτυο δηλαδή αυτό το μέσο. Στόχος είναι να εξοικονομήσουμε χαρτί. Να είμαστε εμείς πρωτοπόροι στην εξοικονόμηση χαρτιού. Κανένας όμως δεν υποχρεώνεται, δεν του το επιβάλλουμε, εκούσια γίνεται για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό εμπειρικά. Και μια συνάντηση τέτοια είχαμε το Δεκέμβριο στο Στρασβούργο και θα υπάρξει και άλλη μια τέτοια συνάντηση τον Ιανουάριο, ώστε οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται και οι βοηθοί όμως επίσης να μπορούν να εξοικειωθούν από αυτό το σεμινάριο όσοι έχουν ενδιαφέρον. Όλοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν. Τρίτη ανακοίνωση, feedback από τον τριμερή διάλογο. Πρώτον το άρθρο 70, εφαρμογή του. Πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Και εδώ η έκθεση ΡΙΣ για παράδειγμα αναφέρεται σε αυτό. Υποδιαπραγμάτευση θέμα και αυτό. Υπάρχει ένα σεμινάριο, workshop για το θέμα της ποιότητας των καυσίμων και με το εργαστήριο που θα έχουμε στις 20 Δεκεμβρίου αυτή την εβδομάδα, 9.30 ώρα και στο κέντρο συνεδριάσεων Αλμπέα Μποσέτ στις Βρυξέλλες. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν πάρει πρόσκληση να παραστούν και συμμετάσχουν. Ε, όσοι θέλουν να παραστούν είναι ευπρόσδεκτοι. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών και 11ης Οκτωβρίου, 5ης και 6 Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις, κυρώνονται τα πρακτικά. Και περνάμε στο σημείο της ημερήσιας διάταξης 4 μετά το 3. Και έχουμε εδώ κάτι, μια έκθεση για τη διάσκεψη των κλιματικών αλλαγών ad hoc στην Τόχα. Είχαμε πάει εκεί με συναδέρφους 15 εκπρόσωποι της Ευρωβουλής ως αντιπροσωπεία πήγαμε στην Τόχα για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και πρέπει να πω, ομολογώ ότι πολλές συνεδριάσεις και συναντήσεις είχαμε με υπουργούς και εκπροσώπους κυβερνήσεων. Ήταν χρήσιμο αυτό και με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Κίνας συζητήσαμε και για τη δική μας νομοθεσία μπορέσαμε να μιλήσουμε για το σύστημα εμπορίας ρήπων, το backloading, αλλά επίσης και όλο τον τομέα των ε, ε, εταιριών ε, εναέριων μεταφορών, εκπομπές ρήπων από τα αεροπλάνα. Ήταν χρήσιμο αυτό και για την αντιπροσωπεία μας που είχε αναφερθεί και το, εστιάστηκε στις τοποθετήσεις όσον αφορά τους εκπροσώπ, τον εκπρόσωπο των Κινέζων για παράδειγμα και συνενετικά θέλουν να εργαστούν οι Κινέζοι μαζί μας, με εμάς τους Ευρωπαίους και αδειμονώ να δω τι θα δώσει το μέλλον από αυτή τη ε, διαδικασία. Αν θα υπάρξει μια ευρεία διεθνή συνένεση τελικά ίσως. Προσπαθήσαμε το δυνατόν περισσότερους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους να συναντήσουμε. Αυτή τη φορά δεν ήταν δυνατόν διότι πολλά εθνικά κοινοβούλια δεν έστειλαν τις αντιπροσωπείες τους στην Τόχα και έτσι το κέντρο βάρους είχε τεθεί σε συναντήσεις με υπουργούς και εκπροσώπους κυβερνήσεων. Εμείς οι ίδιοι είχαμε και μία εκδήλωση που κάναμε που αθρώα την επισκέφθηκαν αυτή την εκδήλωση όπου μιλήσαμε για τη δική μας εμπειρία για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ήταν πλήρης η αίθουσα, μεγάλη συμμετοχή, είχαμε συζητήσεις, είχαμε προσκαλέσει και επαΐοντες τον κύριο Στάινερ για παράδειγμα, τον επικεφαλής του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ και άλλους ε, ειδικού πραγματογνώμενες. Ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο αυτό για την ίδια την διάσκεψη. Πήγαμε την προηγούμενη τελευταία εβδομάδα, από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή. Επίσημο τμήμα που εκτιλήχθηκε τότε. Αλλά οι διασκέψεις αυτές πάνε πάντα στην παράταση και είχαμε εμείς επίσημη εντολή από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή να συμμετάσχουμε εκεί και το πρόγραμμα μας ήταν αρκετά ευρύ, ευρύτατο και κάποια σημεία από το πρόγραμμα επελέγησαν και μέχρι αργά το βράδυ συνεδριάζαμε είτε ωριαία είτε με αναημίωρα και εργαζόμαστε, εργαστήκαμε πολύ καλά και στα σεμινάρια, επιμέρους σεμινάρια, workshops έγιναν υπό την πρωτοκαθεδρία συμμετεχόντων στην αντιπροσωπεία μας. Επικεφαλής ήταν ο, κύριος Καρλ Χάιντς Φλόρενς και εγώ ο ίδιος η ταπεινότητά μου. Πήγαμε λοιπόν στην Τόχα και είχαμε μαζί μας και το ψήφισμα το οποίο είχαμε εγκρίνει ως Ευρωβουλή. Ένα μικρό βήμα ήταν αυτό το οποίο σημειώθηκε όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, όσον αφορά τις προσαρμογές στις κλιματικές αλλαγές. Η μεγάλη απαρχή όμως, η μεγάλη νέα κίνηση δεν μπορούσε να αναμένεται σε αυτή τη διάσκεψη. Σε κάποιους τομείς ε, μάλιστα σε σχέση με αυτές τις ε, με την πρόοδο που μπορούσαμε να σημειώσουμε για τη μακροπρόθεσμη συνεργασία για παράδειγμα και μακροπρόθεσμη δράση το Κιώτο 2 πρωτόκολλο καταφέραμε να το προχωρήσουμε προς έγκριση αυτά δεν είναι πολλά βέβαια και πιστεύω ότι αυτά που εμείς στην Ολομέλεια εγκρίναμε στόχος δύο βαθμών θέρμανσης του πλανήτη και όχι περισσότερο δεν τηρήθηκαν εκεί. Πρέπει κάτι παραπάνω να γίνει λοιπόν. Και αυτό το οποίο σημειώσαμε και παρατηρήσαμε τι ήταν. Στην ίδια την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά από πλευρά των 27 υπουργών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη συντονισμού θέσεων κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε παρουσιάσει με πιο ανάγλυφο τρόπο, με μεγαλύτερη απήχηση, υποσχέσεις για χρηματοδότηση για παράδειγμα, έμεναν ε, μετέωρες. Όταν συναντούσαμε τους ε, κοινοβουλευτικούς μας, εξεπλά, με, με έκπληξη έλεγαν «Μα θα περιμέναμε από τους υπουργούς των 27 ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι παραπάνω». Να μπορούσαν αυτά να παρουσιαστούν στην ε, κοινή γνώμη στους πολίτες και να υπογραμμιστούν περισσότερο. Υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε. Και του χρόνου λοιπόν θα έχουμε και μια τέτοια εκδήλωση και στη Βασοβία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σωστά τα του οίκου της, να εκπονήσει μια στρατηγική ώστε οι επιδόσεις να είναι καλύτερες. Πολλές ανάγκες υπάρχουν που πρέπει να καλύψουμε, μεγάλη πορεία που πρέπει να διανύσουμε. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο το Durban και το μετά το Ντέρμπαν πρέπει να συζητηθούν και στην Ολομέλεια και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Διότι αυτά τα οποία συνέβησαν στην Τόχα δεν πρέπει να επαναληφθούν στη Βασοβία. Πρέπει να προπαρασκευαστούμε πολύ καλά. Και εμεί ω Κοινοβούλιο θα πρέπει με επικριτικό, με κριτικό πνεύμα αλλά και επικοδομητικά να παρακολουθήσουμε και να συνοδεύουμε όλα αυτά. Αλλιώ δεν μπορεί να τηρηθεί και να υπάρξει καν στόχος ε, δύο βαθμών, δηλαδή αναχέτηση σε δύο βαθμούς της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έχουμε πάρα πολλά λοιπόν ε, και πολλούς ε, που έχουν ζητήσει τον λόγο. Ο κύριος Γιώ Λάινεν πρώτος που θα παρέμβει παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την έκθεση της αντιπροσωπείας που δώσατε. Στην Ολομέλεια ούτως ή άλλως θα ξανασυζητήσουμε τα θέματα της Ντόχα. Είπαν κάποιοι, άνοιξε λέει πόρτα για μια νέα εποχή που ξεκινά στην προστασία, παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η αισιόδοξη παραλλαγή. Ίσως άλλοι λένε έκλεισε η πόρτα για την επίτευξη δηλαδή του στόχου της υπερθέρμανσης σε δύο βαθμούς μόνο του πλανήτη. Δεν επετεύχθη αυτό. Είναι στενά τα πράγματα και δύσκολα να σημειωθούν αυτές οι παγκόσμιες πρόοδοι. Δυσχεραίνεται η υπόθεση. Πρέπει φυσικά να διαρωτηθούμε Ποιο ρόλο διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έκανε. Αυτός ο ρόλος είναι ακόμα τόσο καλός και θετικός όπως πριν από κάποια χρόνια ή μήπω έχουμε πολύ λιγότερο λέγειν και πολύ λιγότερο λόγο να αρθρώσουμε και να πούμε κάτι. Σωστό ήταν νομίζω το ψήφισμά μας εμείς να αναφέρουμε την βελτίωση των πραγμάτων με φιλόδοξο στόχο 30% μείωσης. Ούτως ή άλλως θα υπάρξει ανάγκη μέχρι το 2020 να πετύχουμε μείωση όχι κατά 20 αλλά κατά 30% γιατί διαφορετικά το δρομολόγιο μέχρι το 2050 δεν μπορεί να τηρηθεί αν δεν μειώσουμε σε 30% τις εκπομπές ρήπων. Πρέπει να ασκηθεί πίεση τα 30% να εγκριθούν και να θεσπιστούν ως επίσημος στόχος, δεσμευτικός. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κράτησαν οι συμμαχίες που είχαμε στο Ντέρμπαν και με τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, και την ομάδα της καθαγέννηση ε, είχαμε μια ομάδα ως ΕΕ και με τις νησιωτικές χώρες στο Εκεί στην Τόχα δεν είχαμε συμμαχίε. Βρεθήκαμε χωρί συμμάχου. Δεν λειτουργήσαν τα πράγματα όπω αναμέναμε. Και για τη χρηματοδότηση δεν έχουμε να προσφέρουμε τόσα πολλά όσα είχαμε υποσχεθεί στι χώρε. Να πούμε και δύο λόγια για τη ΣΥΠΑ. Όσοι ήταν στην Κοπεχάγη παρόντε θα θυμούνται ότι διαρωτόμαστε τι θα προσφέρει ο Ομπάμα. Και ήταν σαφές ότι δεν είχε τίποτα να προσφέρει ο Ομπάμα γιατί δεν επιθυμούσε το Κογκρέσο. Και έτσι μετά είχαμε μία βαρύγδουπη είδηση 100 δις λέει θα διατεθούν μέχρι το 2020. Δραματική είναι η κατάσταση πρέπει να πω ότι οι ΙΠΑ απουσίαζαν από την Τόχα διότι κάποια τέτοια δέσμευση για 100 δις ε, είναι μετέωρη, δεν είναι καν δεδομένο αυτό είναι κοινική πολιτική. Να λένε 100 δισεκατομμύρια θα τα ρίξουν στην κονίστρα, στο στίβο. Αυτό τι δείχνει. Τεκμηριώνει ότι είναι ανίκανοι και άβουλοι. Δεν θέλουν να μειώσουν τις εκπομπές ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Και δεν θέλουν να συμμετάσχουν προς αυτήν την πορεία. Ο Ομπάμα 2, η δεύτερη θητεία Ομπάμα, πρέπει να προσφέρει πολλά περισσότερα από στο παρελθόν. Αλλιώ θα δυσχερανθεί η υπόθεση πάρα πολύ. Αξιοπρόσεκτη ήταν η ολοκλήρωση και το, η λήξη αυτή. Τη της ε, διάσκεψης. Πώς εγκρίνεται ένα τέτοιο έγγραφο για παράδειγμα όπως αυτό της Δόχα. Εγώ μπορώ να το χαιρετήσω αυτό διότι ελπίζω στο νέο γύρο για τις κλιματικές αλλαγές περισσότερο και καλύτερα από το Κιώτο να μπορεί να υπάρξει μια συνένεση και όχι ομοφωνία. Στο Κανκούν πάλι είχε συμβεί αυτό. η Υπουργοί Εξωτερικών εν μια νυχτή ενέκριναν ένα έγγραφο ενώ η Βολιβία ήταν και εναντίον. Τώρα είχαμε, έχουμε και τη Ρωσία εναντίον. Δεν υπάρχει πρόοδος πιστεύω. Αν αναμένουμε πάντα τον πιο βραδύ οδηπόρο να καλύψει τις αποστάσεις ε, και να προσαρμοστεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μαχιόντας παρακαλώ. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η εργασία μας ήταν αποτελεσματική λόγω της ε, υψηλής ποιότητας της ηγεσία μας. Προσπαθήσαμε βεβαίως μαζί με το Συμβούλιο να μιλήσουμε ε, με μία φωνή και όλοι σεβαστήκαμε το ψήφισμα. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Δεν αποδίδουμε μεγάλη προσοχή τελικά στην επικοινωνία έτσι ώστε δηλαδή να γίνουν γνωστές ε, οι προσπάθειές μας και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά τις εκπομπές. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν που θα ήθελα εγώ να στείλω. Εμείς σαν Επιτροπή Ένβη ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ενεργήσει βάσει των ε, λεγόμενων των επιστημόνων μέχρι το 2020, μείωση λοιπόν κατά 5% των εκπομπών. Αλλά εάν δεν συμφωνήσουν σε αυτό και οι άλλοι μας εταίροι, τότε όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, αλλά τελικά θα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα χαθούν θέσεις απασχόλησης και στην ουσία θα κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Επομένως, ε, ε, οι διαπραγματεύσεις ε, καταδεικνύουν σαφώς ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην κινητήρια δράση που πρέπει να έχει η πολιτική μας. Θα πρέπει οι πολιτικές μας να είναι και πιο δραστήριες και πιο φιλόδοξες. Τελευταίο μήνυμα. Το υλικό μας ε, το προετοιμάσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό και τη Γραμματεία και όλους όσους μας βοήθησαν στη διάρκεια αυτής της αντιπροσώπευσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφε για όσα είπατε και σε σχέση με την Ελίσαβεθ και τον Ιωσέφ που πασκεύασαν εξαιρετικά αυτό το θέμα, πάντα μα οδήγησαν με ασφάλεια. Είχαν παρασκευαστεί όλα τέλεια. Σε μια τέτοια διάσκεψη, αν υπάρχουν απρόβλεπτα θέματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Έπαινο, υψηλό έπαινο σε αυτούς τους δύο και σε του άλλους συμμετείχαν για την εξαιρετική επίδοση. Στη συνέχεια, ο Επαΐων που είναι και πραγματικά ο Κρήτον Ασένη επαίων για τα θέματα αυτά στην Τόχα. Κύριε Ασένη, έχετε τον λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω και εγώ ε, και υπογραμμίζω ότι όλοι ήταν ε, με φθόνο κοιτούσαν αυτό το βιβλιαράκι που είχαμε, που μας είχε προετοιμάσει η γραμματεία. Επομένως ε, και εγώ ευχαριστώ τη γραμματεία για τη δουλειά. Είχαμε καλά νέα και κακά νέα από την Τόχα. Τα καλά νέα είναι ότι έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις. Προχωράει ο κόσμος έτσι ώστε ε, να συμφωνήσει, αλλά τα κακά νέα είναι ότι είναι πάρα πολύ αργός ο ρυθμός ε, αυτής ε, της ε, πρόοδου. Έτσι, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να είμαστε στο ραντεβού του 2050 με μια νέα, συγγνώμη, 2015, μέχρι, έτσι ώστε να έχουμε μέχρι τότε δηλαδή μια, ένα συμφωνημένο κείμενο με συμφωνημένες αρχές. Ε, θα πρέπει ο καθένας, ε, η κάθε χώρα προετοιμάζει ε, την κατάσταση βάσει της εντολής της διαπραγματικής που έχει και πραγματικά σας λέω ότι με μεγάλη δυσκολία πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τη συμφωνία μέχρι το 2015. Αυτό σημαίνει πολλά και για το Κοινοβούλιο έχουμε ευκαιρίες στο Κοινοβούλιο για να δράσουμε με διαφορετικό τρόπο, για να βοηθήσουμε, για να συμβάλλουμε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει διαφορετική, διαφορετικός τρόπος δράσης και στα ευρωπαϊκά όργανα. Αλλά μέχρι τώρα υποβάλαμε ψηφίσματα ε, πρώτης ε, διασκέψεως κορυφής ε, του Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Of the, of the uh, run, which was a marathon, but now it's... Και μέχρι τώρα είχαμε μαραθώνιο, αλλά τώρα θα πρέπει να βρεθούμε στο τελικό σπριν των 100 μέτρων. Επομένως, αν είναι δυνατόν, πρέπει να προετοιμάζουμε ψηφίσματα και για τις ενδιάμεσες ε, συναντήσεις. Έχουμε άλλη μία συνάντηση στην Βόνη. Θα πρέπει από κοντά να παρακολουθούμε, να βλέπουμε τι γίνεται. Ένα πολύ στενό monitoring λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε όποτε αυτό είναι απαραίτητο γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Εάν οι χώρες δεν αυξήσουν την φιλοδοξία τους όσον αφορά τις διεθνείς τους θέσεις και αν δεν διευρυνθεί και η διαπραγματευτική εντολή, όποια ψηφίσματα και αν εκδίδουμε εμείς ε, θα φτάνουν πάντα πολύ αργοπορημένα, ε, θα δείχνουν έτσι μία υπεραισιόδοξη άποψη για τις ε, διαπραγματεύσεις γιατί τελικά η κάθε μία χώρα θα χρειάζεται το χρόνο της έτσι ώστε να, κάνει, να προετοιμάσει τη διαπραγματευτική εντολή. Επομένως να είμαστε έτοιμοι σε εθνικό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε γρήγορα ε, στην, ε, στην τελική συμφωνία. Μεγάλη, μεγαλύτερη λοιπόν φιλοδοξία, μεγαλύτερο βάρος στις διαπραγματεύσεις, ετοιμότητα έτσι ώστε ε, να είμαστε έτοιμοι σε κάθε θητεία να παρεμβαίνουμε. Όταν μιλάμε για θέσεις εθνικών αντιπροσωπιών, να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι έτοιμες να πράξουν με τον ίδιο τρόπο. Κυρία Ρεπάζ, παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και εσάς ε, για την καθοδήγηση αυτής της αντιπροσωπείας και τη γραμματεία για την προετοιμασία της. Την εξαιρετικά καλή προετοιμασία της. Θα συμφωνήσω με τις πρότασεις Γιολάινεν. Ε, παρακολουθώντας τις συνόδους μετά την Κοπενχάγη, η σύνοδος που έλαβε χώρα στη Ντόχα σήμανε, πιστεύω, αποδυνάμωση της θέσης της Ευρώπης σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το συζητήσαμε εξάλλου πολλέ φορέ μεταξύ μα υπήρξαμε υπερβολικά και εδώ θα χρησιμοποιήσω λίγο έντονα λόγια μας έκριναν υπερβολικά τόσο οι χώρες του Νότου όσο και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ενώ εμείς σήμερα είμαστε η μόνη περιοχή του κόσμου που έχουμε δεχθεί μαζί με την Αυστραλία, την Ελβετία και την Νορβηγία φυσικά αλλά τελικά δεσμευτικές ε, υποχρεώσεις ε, όπου έχουμε προτείνει χρηματοδότηση για την περίοδο 2013-2014 και πραγματικά κάνουμε προσπάθειες πιο σημαντικές. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αξιόπαινες, αξιόπαινες προσπάθειες. Και παρόλα αυτά μας επέκριναν διάφορες χώρες, όπως και η χώρα που μας υποδέχτηκε, το οποίο είναι απολύτως παράδοξο. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιους προβληματισμούς. Όσον αφορά τις διπλωματικές κινήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά τη Σύνοδο για το κλίμα και γενικότερα για το θέμα ε, ενώπιον των εταίρων μας είτε εταίροι από βιομηχανοποιημένες χώρες είτε από χώρες του Νότου είτε πρόκειται για μη κυβερνητικούς οργανισμούς ώστε να αναδείξουμε καλύτερα την αξία των όσων κάνουμε και να μπορούμε να προλάβουμε τις ε, ενδεχόμενες κριτικές που μπορεί να διατυπωθούν. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή παράδοξο. Ότι αυτά τα πολύ μέτρια αποτελέσματα της Συνόδου της Ντόχα όσον αφορά τα διαφορετική βεύματα δεν πρέπει να θέτουν στην άκρη τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου και εγώ έχω την αίσθηση και δεν ξέρω αν όλοι έχουν την ίδια αίσθηση όσοι παρέστησαν στην Ντόχα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ότι απομακρυνόμαστε από μια διεθνή διακυβέρνηση σε κλιματικά θέματα και κινούμαστε περισσότερο προς τη σπουδαιότητα των εγχώριων μέτρων. Ας δούμε τι μας είπε η κινέζικη κυβέρνηση, τι μας είπαν οι Ιάπωνες, τι κάνει η Κορέα, τι κάνουν πολλές άλλες χώρες. Κοιτάζοντας όλα αυτά, καθίσταται σαφές ότι οι υπερβολικά φιλόδοξες πολιτικές υλοποιούνται σε διάφορες χώρες του κόσμου Παρόλα αυτά δεν καταλήγουμε σε καλά αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνούς διακυβέρνησης. Υπογραμμίζω λοιπόν το λάθος που θα κάναμε ως Ευρωπαίοι αν νομίζαμε ότι επειδή δεν προχωράμε σε επίπεδο διεθνούς διακυβέρνησης σε κλιματικά θέματα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε ενδιαφέρον για επενδύσεις και φιλόδοξες πολιτικές ε, στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας, διότι οι υπόλοιπε χώρες επενδύουν πολύ. Εάν λοιπόν εμείς δεν δραστηριοποιηθούμε έντονα σε αυτούς τους τομείς, ε, θα χάσουμε ε, τόσο από πολιτική άποψη επειδή είμαστε ηγέτες σε αυτό το θέμα, αλλά θα χάσουμε επίσης και πολλά σε βιομηχανικό και οικονομικό μέτωπο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το ότι πηγαίνουμε αργά σε διεθνές επίπεδο δεν σημαίνει ότι ε, αργοπορούν τα κράτη σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τι βιομηχανικέ και οικονομικέ πολιτικέ που υλοποιούνται. Κυρία Όλσκοκ, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και όλους τους υπόλοιπους για την άριστη δουλειά τους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ντόχα. Θα συμφωνήσω με την Κορίν Λαπάζ. Και εγώ ήμουν παρούσα στις τέσσερις συνόδους για το κλίμα και καθίσταται απολύτως αφές πώς ε, ο κοινός τόπος που είχαμε αρχίζει να ε, χωρίζεται σε διάφορα μέτωπα. Υπήρχαν πολύ φιλόδεξες χώρες όπως η Νορβηγία. Αλλά πολλές άλλες χώρες, η Κίνα έχει φιλοδοξίες δικές της, αλλού τύπου και υπάρχουν και ευρωπαϊκές χώρες με, με πολλές φιλοδοξίες. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, Τελικά μιλάμε για μια ανοιχτή ε, σύνοδο ουσιαστικά διερεύνησης κεφαλαίων, αναζήτησης κεφαλαίων ε, για φιλανθρωπικούς σκοπούς ας πούμε όπου η κάθε χώρα δίνει ό,τι πιστεύει ότι μπορεί να δώσει στο καλάθι συνεισφέρει όπως μπορεί απλά για να το δείξει στους ψηφοφόρους στις χώρες τους. Αυτό μπορούμε να το επιτρέψουμε να γίνει για μια μεταβατική περίοδο, αλλά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μάλλον θα πρέπει να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση ε, ενοποιημένου μετόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η, συνεδρία, η διαφορά μεταξύ της προηγούμενης συνόδου και αυτής. Διότι τότε μιλούσαμε για το αποτέλεσμα των συζητήσεων και αναφέρθηκε ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση του Κοινοβουλίου, της Κομισιόν. Ε, βρισκόμασταν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ενώ αυτή τη φορά ήμασταν χωρισμένοι θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε αυτό, να μας προβληματίσει. Όπως είπατε στην αρχή, εγώ θα έλεγα ότι παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξη. Διότι παρότι αυτή η συνάντηση, η σύνοδος ήταν μάλλον βασίστηκε σε ό,τι μπορέσαμε να αυτοσχεδιάσουμε επί τόπου τελικά ορισμένες φορές καταλήγει κανείς σε μια κατάσταση όπου όλος ο κόσμος βρίσκεται σε οικονομική κρίση και παρόλα αυτά καταφέραμε καταφέραμε να επιτύχουμε ορισμένα πράγματα σε ουσιώδη θέματα αλλά χρειάζεται να σημειωθεί πρόοδος στην επόμενη σύνοδο αλλά χρειαζόμαστε κάποιο ανοιχτό δίκτυο, ανοιχτό προς όλους, όλου όσου συμμετέχουν σε συνόδους για το κλίμα, όσου έχουν συμμετάσχει και που έχουν δεσμευτεί ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι πρέπει να προετοιμαζόμαστε και μεταξύ των, στο εσωτερικό των συνόδων και μεταξύ δύο συνόδων δεν λέω ότι πρέπει να ανταγωνιζόμαστε την Κομισιόν αλλά να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων με τους οποίους συναντιόμαστε, με τους οποίους συνεργαζόμαστε καθημερινά και πιστεύω ότι θα χρειαστεί να επιταχύνουμε και να ανεβάσουμε λιγάκι τα στάνταρ μας. Έχουμε τη συνάντηση στη Βόνη την Άνοιξη και μετά τη συνάντηση στη Βαρσοβία. Και δεν πρέπει να αφήσουμε να, να, να θεωρηθεί ότι βάζουμε τροχοπέδι συνέχεια. Θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε φυσικά είναι σημαντικέ και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να κάνουν πολύ καλή εντύπωση σε αυτέ τι συνόδου. σω την επόμενη φορά να υπάρξει ένας προϋπολογισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, το Κογκρέσο ίσως να είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τον πρόεδρο που βρίσκεται στο μέσο της τελευταίας του θητείας. Δεν μπορεί να επανεκλεγεί. Πιστεύω ότι εντό τη κυβέρνηση Ομπάμα έχει εκφραστεί τεράστια δέσμευση για τα κλιματικά ζητήματα. πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο. Όχι να είμαστε αδύναμοι. Σα ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο αγορητών και έχουμε και την Επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που έχουμε εκπρόσωπό τη. Παρότι, την, παρόλη τη μεγάλη ανάγκη συντονισμών και διαπραγματεύσεων υπήρχε χρόνος για την αντιπροσωπεία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο με μια ενημέρωση επικαιροποιημένη όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Καλοχαιρετίζω τον επικεφαλής διαπραγματευτών για την Επιτροπή στην Τόχα που ήταν παρόν, τον κύριο Αρτούρ Μέτσκε. Παρακαλώ, έχει κύριε Μέτσκε τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και βεβαίως ήταν μεγάλη χαρά και για μένα να ε, είμαι στο ίδιο ε, σημείο με το Κοινοβούλιο και κυρίως να μην έχουμε ανταγωνιστική σχέση με το Κοινοβούλιο όπως άλλωστε σημειώθηκε ήδη. Θέλαμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και το επιθυμούμε ακόμα. Πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε που μας ε, περιμένουν. Θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη, στον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης το 2015 ε, στο Παρίσι. Αλλά βεβαίως εντωμεταξύ έχουμε και τη Βαρσοβία του χρόνου. Ε, και επομένως πολλή δουλειά έχουμε σαν Ευρωπαίοι. Πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως καμιά φορά όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, καμιά φορά έτσι έχουμε ε, περισσότερες φιλοδοξίες ε, ή ε, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Όχι, και στην Κοπενχάγη και στα Κανκούν καταφέραμε κάποια πράγματα και αυτά που πετύχαμε εφαρμόζονται ήδη ενώ, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και το, στο μέλλον και έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά και να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, για την αλλαγή του κλίματος. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν αλλά διστάζουν ε, και να δεσμευτούν σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πρέπει να αλλάξει τα επόμενα χρόνια γιατί ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας πέρα από το 2020 δεν θα είναι εύκολος, μάλλον θα είναι λίγο πιο δύσκολος δύσκολες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν, δύσκολα πράγματα μας περιμένουμε. Μιλάμε για ευθυνή ενέργεια, μιλάμε για ενεργειακή ε, αυτάρκεια και ενεργειακή αποδοτικότητα. Όλα αυτά μας περιμένουν στη στροφή του 2020 και επομένως θα πρέπει όλοι να δουλέψουν λίγο πιο πολύ από ό,τι πιστεύαμε πριν την Κοπεχάγη. Το δεύτερο που θέλω να πω όσον αφορά την φιλοδοξία των στόχων, ναι, ε, νομίζω ότι και στην Τόχα για μία ακόμα φορά αναγνωρίστηκε ότι εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε κάτω από τους δύο ε, βαθμούς, αλλά όλοι αναγνώρισαν ότι το 2013 ε, και 2014 συμφωνήθηκε να γίνει επιπλέον προσπάθεια έτσι ώστε να δουν τα εμπλεκόμενα μέρη τι μπορούν να κάνουν μέχρι το 2020 και ε, σε το 2014 στη συνάντηση υπουργικού επίπεδου να συζητηθεί ακριβώς αυτό είναι σωστό ότι ε, τα στοιχεία που θα βάλει στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, τα μάλλα εξαρτώνται από αυτά τα οποία θα αποφασιστούν στο Συμβούλιο του επόμενου 18 μήνες. Υπάρχει πρόταση και από την ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πάρα πολλά θέματα, για διαρθρωτικά μέτρα, για την, τον έλεγχο των ρήπων, των εκπομπών κτλ. Όλα αυτά συζητιούνται. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά για, για τον καθορισμό της διαπραγματευτικής θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα δύο χρόνια. Τρίτον, το ζήτημα της, των αποφάσεων στην Τόχα. Είναι ορθόν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, εκπροσωπώντας όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και την Ουκρανία και την Λευκορωσία, στην τελική ολομέλεια, ήταν κατά της ε, απόφασης όσον αφορά την δεύτερη περίοδο δέσμευσης. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον προσπάθεια έτσι ώστε να ξαναφέρουμε και την Ουκρανία και την ε, Ρωσική Ομοσπονδία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί εάν το 2015 έχουμε συμφωνία χωρίς τις δύο αυτές χώρες, ε, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους ανταγωνισμό ακριβώς στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εμπλακούν στη Συμφωνία του 2015. Δεν μπορεί να γίνει η Συμφωνία του 2015 χωρίς αυτές τις δύο χώρες. Ε, μία τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω όσον αφορά την συμμαχία με τις λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες και με τους προοδευτικούς Λατινοαμερικανούς είναι ορθό ότι αυτή η συμμαχία δεν ήταν τόσο εύκολη όσο στον Τέρμπαν. Και όσον αφορά τη δεύτερη ε, περίοδο δέσμευση, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Είπαμε λοιπόν ότι ε, οι χώρε οι οποίες ε, θέλουν να πάνε σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, αυτοί θα εξαρτώνται περισσότερο από εμά. Κυρίως όταν μιλάμε για μικρές νησιωτικές χώρε, μικρά νησιά, τις λιγότερο αναπτυγμένε περιοχές ε, προκύπτουν ε, ζητήματα. Πάντως πρέπει να πω ότι ο τόνος των διαπραγματεύσεων άλλαξε άρδινε τη δεύτερη εβδομάδα. Έγινε περισσότερο πολιτική στάση και λιγότερο τεχνοκρατική. Και πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε έτσι, ε, αυτά τα προβλήματα στις επαφές που έχουμε με τις χώρες αυτές και εν τέλει να ε, υπερκεραστούν τα εμπόδια. Έτσι, το σημαντικό είναι ότι ε, συνεχίζεται η συζήτηση έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο το επίπεδο των φιλοδοξιών όχι μόνο μετά το 2020 αλλά και πριν το 2020 και μπορούμε να στηριζόμαστε σε αυτή την συμμαχία τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, κυρίως όσον αφορά ε, την χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή, όταν δηλαδή θα αρχίσει να λειτουργεί και το ε, ταμείο, το πράσινο ταμείο και μετά το 2020 βεβαίως όταν θα μπορούμε να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία και για τους συμμάχους μας και για, την χώρα, για τις χώρες της Αφρικής. Σας ευχαριστούμε κύριε Χωνεμέτσκα. Ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση για αυτή την έκθεση για την αντιπροσωπεία μας και θα πρέπει το μπαλάκι να το λάβουν και να δοθεί συνέχεια ώστε διαρθρωτικά, δομικά να εξετάζουμε αυτά τα προβλήματα όχι μόνο πριν από τις διασκέψεις αλλά και ενδιάμεσα και να προβληματιστούμε να δούμε ποια στρατηγική το 2013 θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να καταλήξουμε και το 2014 στο Παρίσι και όσον αφορά και την κοινωνία των πολιτών το θέμα αυτό δεν ήταν απόλυτα παρόν στις πρώτες σελίδες ε, των μέσων ενημέρωσης. Κάτι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τονίσουμε την αναγκαιότητα να γίνει αυτό και στα κράτη τα κράτη-μέλη από τα οποία προερχόμαστε να μεριμνήσουμε αυτό να αναβαθμιστεί στην ημερήσια διάταξη, να έχει προτεραιότητα όσον αφορά τα άλλα θέματα και να μην αγνοείται, να μην αμελείται. Ευχαριστώ. Αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία και για την πιθανή προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και την προώθηση αυτού του θέματος. Έτσι. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και εδώ τι έχουμε. Θεματολογικά ταιριάζει πολύ καλά αυτό με το προηγούμενο, γιατί είναι κάτι πολύ χειροπιαστό και συγκεκριμένο. Να πετύχουμε τους στόχους για τις αλλαγές, τις κλιματικές αλλαγές και σε παγκόσμιο επίπεδο, διεθνώς, να δείξουμε ότι έχουμε σοβαρές προθέσεις με την καταπολέμηση των ε, κλιματικών αλλαγών. Το πιο δυνατό μέσο μας είναι το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων. Πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό, πώς μπορεί να λειτουργήσει και να είμαστε πιο αποδοτικοί, να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και σε σχέση με το 2003-87 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την διευκρίνηση διατάξεων που αφορούν τα χρονοδιαγράμματα πληστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Βρισκόμαστε στην τρίτη περίοδο δράσης που ξεκινά από την 1η Πρώτου 2013. Κατά τη διάρκεια του, πακέτου για το κλίμα και τις εκπομπές ρήπων, αποφασίσαμε πώς θα πρέπει, πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτά και υπήρξαν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια μορφή θα πάρουν αυτές οι προτάσεις και υπήρξαν αποφάσεις. Θυμάμαι πολύ καλά μια τέτοια απόφαση, την απόφαση για τα CDMs που είχαμε τότε εγκρίνει στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Αμέσως μετά την ψηφοφορία είχα πολύ μεγάλα προβλήματα και διαρωτήθηκα, θα είχαμε ευκαιρία, έχουμε ευκαιρία ως Ευρωκοινοβούλιο αυτή την αγορά των CDMs να αποφύγουμε να πλημμυριστεί, να υπάρξει μια πλημμυρίδα με τέτοια πιστοποιητικά. Διαπιστώθηκε ότι είχαμε μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και έτσι η παραγωγή δεν αυξήθηκε περαιτέρω, αλλά αποτελματώθηκε λίμνασε η παραγωγή, έμεινε στάσιμη και έχουμε πάρα πολλά, υπερβολικά πολλά πιστοποιητικά διοξιδίου του άνθρακα στην αγορά. 955 εκατομμύρια τέτοια πιστοποιητικά που κυκλοφορούν στις αγορές. Αύξηση αυτό δηλαδή και η τιμή του κάθε πιστοποιητικού είναι 7 ή 8 ευρώ ανάλογα <clears throat> με το πώς βρίσκεται η κατάσταση, αν ακολουθεί αυξητική ή φθήνουσα πορεία. Και όταν τότε συζητήσαμε αυτό το πακέτο μέτρων, αυτή τη δέσμη μέτρων, ο πύχης ήταν, ο γνώμονας, είχε τεθεί στα 30 ευρώ. Και όχι σε αυτές τις χαμηλές τιμές. Βλέπουμε σε αυτές τις τιμές που έχουμε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια δεν αυξάνονται, δεν βελτιώνονται οι επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες. Αν το αντίθετο έχουμε επενδύσεις και σε σταθμούς ε, παραγωγής ηλεκτρικού, ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Και δεν μπορεί αυτό μακροπρόθεσμα να θεωρείται κάτι το οικονομικό και θετικό. Κατά τούτο λοιπόν παρενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρενέβη και λίγο πριν από τις θερινές διακοπές υπέβαλε μια πρόταση για το αποκαλούμενο backloading. Δηλαδή, πιστοποιητικά θα πρέπει να αφαιρεθούν, να αποσυρθούν από την αγορά. Είχα την τιμή εγώ να παρακολουθήσω την έκθεση στην Ευρωβουλή. Αυτή ήταν η επιθυμία των συντονιστών θα έπρεπε από πλευρά ε, Προεδρία ε, Επιτροπή, Προέδρου Επιτροπή να μπορέσει να προχωρήσει. Ήταν πολύ σύντομη αυτή η έκθεση, αυτή η γνωμοδότηση. Το μόνο που θέλαμε είναι να δημιουργηθεί νομική βεβαιότητα, νομική ασφάλεια. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, το τολμούσε και υπέβαλε αυτή την πρόταση, αυτά τα πιστοποιητικά να αφαιρεθούν, να αποσυρθούν από την αγορά. Στην Επιτροπή για τα θέματα τα κλιματικά, των κλιματικών αλλαγών συζητώνται αυτά για μένα ήταν σημαντικό. Δεν είχαμε μια πραγματική ακρόαση, αλλά μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος γι' αυτό. Και αυτά τα οποία εγώ <clears throat> είδα και μεριμνήσαμε να γίνουν είναι <clears throat> αυτή η διαδικασία άπαξ να μπορεί να λειτουργήσει και να μην γίνει μια μόνιμη διεργασία, διαδικασία. Αυτά όλα περιέγραψα στην έκθεσή μου μία τέτοια παρέμβαση να γίνει. Και ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφέ και αυτό το συμπεριέλαβα. Αυτό δεν είναι λύση του προβλήματος. Αναβάλουμε τη λύση του προβλήματος χρονικά. Μεταθέτουμε χρονικά την αντιμετώπιση. Διότι αφαιρούνται από την αγορά κάποια πράγματα τα οποία μετά μπορεί να επανέλθουν. Δηλαδή, αεφέτος θα πρέπει οι χώρες να δουν πώς αυτό το σύστημα θα διαμορφωθεί και θα καθοριστεί για το μέλλον και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σχέση με τους πολίτες για ένα τέτοιο, για αυτό το σύστημα. Διότι είναι σαφές και στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης κάνουμε λόγο για εκπομπές ρήπων και για εναέριες μεταφορές αν όλα τα 27 κράτη-μέλη όπως οι συμμετέχοντες από την Ιαπωνία μας είπαν στην Τόχα θεσπίσουν και εισαγάγουν τέλη για το ε, διοξίδιο του άνθρακα θα υπάρχει στρέβλωση στην αγορά. Γι' αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας. Έχουμε κάθε συμφέρον οι εκπομπές ρήπων να διαμορφωθούν σε ένα συνετό λογικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αδειμονώ και προσβλέπω να δω πώς θα διαμορφωθεί η συζήτηση και τι θα πούν οι αρμόδιοι. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο περί του οποίου πρόκειται είναι το backloading να αντιμετωπιστεί και να δράσουμε. Δεν θέλουμε το σύνολο του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρήπων να το αναδιαρθρώσουμε, να το συζητήσουμε, δεν θα έφτανε και το χρονικό πλαίσιο. Έχουμε κάθε συμφερόν των δυνατόν λιγότερες αλλαγές και τροποποιήσεις να υποβληθούν, να ενταχθούν σε αυτή τη διεργασία. Και η δομημένη, διαθρωμένη συζήτηση να διεξαχθεί σε άλλο σημείο, εκεί όπου πρέπει να γίνει και εκεί όπου θα έχουμε και αρκετό χρόνο, επαρκή χρόνο να διεξαγάγουμε μια τέτοια εμβαθυμένη συζήτηση. Και με την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να δοθεί δοθεί μια επισήμανση σε αυτήν ποιε είναι οι απόψει του Ευρωκοινοβουλίου. Τι θέλουμε να γίνει με τι εκπομπέ λοιπόν. Εδώ με το backloading λοιπόν μόνο χρόνο εξαγοράζουμε. Μεταθέτουμε την επίλυση του προβλήματο μεταγενέστερα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Και το συμφέρον μα είναι η έκθεση αυτή να συζητηθεί το δυνατόν καλύτερα και σε μεγάλο βάθο και το χρονοδιάγραμμα το έχουμε καθορίσει έτσι ώστε να μην πάμε πολύ βιαστικά καλπάζοντας, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα νυφαλιότερα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα αναμεταξύ μας. Αλλά το δυνατόν με λιγότερες τροπολογίες και αλλαγές και τροποποιήσεις, ώστε να μπορέσουμε μέσα στο χρόνο που θα έχουμε το δυνατόν πιο γοργά αυτό το backloading να το νομιμοποιήσουμε από την Ευρωβουλή, να το θεμητοποιήσουμε και να προχωρήσουμε γοργά. Απευθύνουμε προς το Συμβούλιο. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. εμεί εδώ να κάνουμε τα του οίκου μας, τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και να είμαστε εντάξει και στο Συμβούλιο η συζήτηση αυτή να αναβάλλεται εσαΐ επαόριστον και στο τέλος οι 27 Υπουργοί να μην κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να συμφωνήσουν <clears throat> ότι θα πρέπει η συζήτηση για την έκθεση για την αγορά ε, ε, εκπομπών ε, ρήπων για τον άνθρακα θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση. Αυτή είναι μια έκκληση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος γιατί διαφορετικά η συγκυρία θα είναι αρνητική από πλευρά των Υπουργών Περιβάλλοντος και δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Εμείς θέλουμε το δυνατόν πιο γοργά η πολιτική για το περιβάλλον να διαμορφωθεί και να καθοριστεί από εμά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσει τα επόμενα χρόνια να λειτουργήσει αντισταθμιστικά για να βελτιωθούν τα πράγματα. Διαφορετικά θα έβαιναν τα πράγματα κακώ και για την αξιοπιστία μα αλλά και για την προστασία του κλίματο και για τι μελλοντικέ διασκέψει για το κλίμα. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια και θα πάμε με τη σειρά στους όσους θέλουν να λάβουν ο λόγο και όδη συγητέ με τη σειρά. Πρώτη, η συνάδελφο Κόρολα. Παρακαλώ. Yes, thank you very much. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για την εργασία του που οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά που δεν είναι αρκετά μεγάλο βήμα. Η έκθεση κάνει αυτό που θέλει η Κομισιόν και μόνο δηλαδή να βγουν οι άδειε από την αγορά. Η Κομισιόν διαρκώς αναφέρει ότι ε, θα πρέπει τα δικαιώματα από την αγορά ε, ε, και η Κομισιόν διαρκώς το λέει αυτό. Εδώ θέλαμε αυτό να δημιουργήσουμε σαν ένα νέο εργαλείο ε, για την αγορά, το οποίο θα το διαχειριζόμαστε ε, με σωστό τρόπο σε σχέση, ε, στη σχέση κόστους ωφέλους και ότι θα βοηθήσει την βιομηχανία. Φαίνεται όμως ότι ο χειρότερος εχθρός του ETS είναι η ίδια η Κομισιόν και τελικά φαίνεται ότι είναι η ίδια η οποία αντιτίθεται στη δημιουργία, την πραγματική δημιουργία της ελεύθερης αγοράς ενέργειας. Η ίδια καταλαβαίνει είναι βεβαίως ότι προσπαθεί λίγο να βελτιώσει την κατάσταση έτσι ώστε να έρθει ε, να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά. Όμως ε, με αυτά τα πισωγυρίσματα τελικά δημιουργεί σύγχυση ε, η οποία προκύπτει από την μεγάλη ασάφεια και την μεγάλη αβεβαιότητα που δημιουργείται. Ε, είναι γεγονός ε, ότι ε, αυτό που λέει η Κομισιόν, ότι η τιμή αυτή τη στιγμή είναι χαμηλά, αλλά ας μην κρύβεται πίσω από το δαχτυλό της η Κομισιόν, θα δει ότι υπάρχει ύφεση παντού και ότι γενικώ υπάρχει μια πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά την ενέργεια και την αποδοτικότητα της ενέργειας. Η Κομισιόν θα πρέπει τώρα να εστιάσει τις προσπάθειές της ε, μαζί με τις προσπάθειες των κρατών μελών έτσι ώστε το σύστημα αυτό να γίνει ε, πιο αποδοτικό και εν πάση περιπτώσει να μπορεί ε, να δίνει ενέργεια στους καταναλωτές σε όχι πάρα πολύ υψηλή τιμή. το, από, το 2000, ε, το 2020 στο 2022 φτάσαμε για τους ε, στόχους ε, και τελικά αυτό το εργαλείο δημιουργείται μονάχα για να, δημιουργούν, για να δημιουργούνται ας πούμε κάποιες νέες χρεώσεις δήθεν για την ενσωμάτωση του κόστους των ανανεώσιμων ποιών ενέργειας και τώρα ε, φαίνεται ότι θέλουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την τιμή. Αναρωτιέμαι όμως, τι την απασχολεί πιο πολύ την Κομισιόν, το, η λειτουργία του ETS ή η λειτουργία ε, της ε, οικονομίας μας και της κοινωνίας μας εν τέλει. Αυξάνεται το κόστος της ενέργειας με αυτούς τους τρόπους και θα υποφέρουν όλοι με την ε, προτινόμενη τροποποίηση του συστήματος δημοπρασιών και του χρόνου μάλλον των δημοπρασιών δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν απλώς ε, να ε, εξακολουθήσουμε την ίδια γραμμή όσον αφορά το ETS και τελικά να μην εξυπηρετούμε αυτούς για τους οποίους αρχικά δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην ε, οικονομική ανάκαμψη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην, στην μη δυναμίτηση του ιδίου, της ιδίας αρχής του συστήματος ε, ETS οι μεγαλύτεροι χρήστες ε, του ηλεκτρικού, της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μπορεί να δουν διπλασιασμό, βλέπετε τριπλασιασμό της ενεργειακής ε, του ενεργειακού τους κόστου στα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή και οι προτινόμενες τροποποιήσεις ε, των δημοπρασιών αντιτίθενται στο ETS. Ε, στο άρθρο 9 απαγορεύεται ας πούμε οποιοδήποτε backloading από τη μία χρονιά στην άλλη. Αυτή είναι πολύ συσταλτική ερμηνεία όσον αφορά την ποσότητα και το μέγεθος των δικαιωμάτων. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε υποτίθεται έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ε, το σύστημα να είναι προβλέψιμο και η ίδια η Κομισιόν είναι αυτή η οποία υποβαθμίζει και δυναμητίζει το σύστημα αυτό ε, και αλλάζει τον τρόπο δημοπράτησης και τον τρόπο κατανομής. Το άρθρο 9 όμως είναι σαφές και επομένως ε, προφανώς δεν θα αρκεί μια τροποποιητική τροπολογία έτσι ώστε να αλλάξει η θέση της ε, Κομισιόν η οποία φαίνεται ότι διαβάζει με τελείως διαφορετικό τρόπο το άρθρο 9. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε να ενσωματωθούν όλα αυτά στην τιμή της ενέργειας μετά το 2020 διατηρώντας όμως και τον, την ανταγωνιστικότητά μας. Σας ευχαριστούμε κυρία Κόρολα. Όχι, Ντέβις, ποιος. Εσείς ούτε Βίλα εδώ. Μάρτιν Κέλλερ δεν παρίσταται. Σαμπίνε. Ωραία, εντάξει. Άννα Χάσμαχ, παρακαλώ. Ο νέος Μάρτιν, έχετε τον λόγο, παρακαλώ Άννα. Sorry, Oh, thanks a million. That's most kind of you. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας μου ζήτησε, επειδή έχει καθυστερήσει το τρένο του, μου ζήτησε να διαβάσω τη δήλωσή του. Το ETS έπρεπε να βασίζεται στην αγορά ως μηχανισμός ώστε να αποφασίζονται οι τιμές βάσει της ζήτησης τελικά. Σήμερα μας λένε ότι η αγορά ανθρακούχων εκπομπών δεν είναι φυσιολογική αγορά. Αληθεύει αυτό, διότι δημιουργήθηκε τεχνητά εμείς όμως συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να βασίζεται σε κανόνες της αγοράς και ότι θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την απόφαση. Σε εποχές οικονομικής κρίσης θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουμε αποφάσεις οι οποίες ενδέχεται να επιβαρυνούν τη βιομηχανία. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι το πλεόνασμα των δικαιωμάτων οφείλεται σε αυτή την κρίση και στις χαμηλότερες, στα χαμηλότερα ποσοστά παραγωγής. Το να αφαιρέσουμε μια ποσότητα έστω και προσωρινά δικαιωμάτων από την αγορά μπορεί να βοηθήσει την ανάκαμψη. Εφόσον αναμένουμε οικονομική ανάκαμψη, είναι αδύνατο να προβλέψουμε τις τιμές επειδή ο μηχανισμός της αγοράς θα επηρεάσει και αυτές. Συνεπώς, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε υπόθεση κάνει η Κομισιόν για να επηρεάσει τον backloading των τρέχουσων τιμών είναι απολύτως αβέβαια. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα πράγματα που με ανησυχούν Τι σημαίνει σωστή λειτουργία της αγοράς μετάξε. Από αυτή την άποψη η πρόταση του εισηγητή μπορεί να, να αποτελέσει μια καλή, ένα καλό σημείο αφετηρίας για να καθοριστεί τι εξουσίες θα λάβει η Κομισιόν. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το κομμάτι αυτής της έκθεσης, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την άλλη υπόθεση, το άλλο σενάριο που προβάλλει ο εισηγητής για ότι πρέπει να ακολουθήσει πιο βαθιά αλλαγή στο σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανά ο συνάδελφος Θαδέος Σιμάνσκι έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση για αυτό το θέμα που αυτή τη στιγμή διεξάγεται δεν μπορεί να διαχωριστεί αυτή η συζήτηση όσον αφορά τις, τους συνολικούς συσχετισμούς μεταξύ θεμάτων για τη διάσκεψη για το κλίμα μόλις ακούσαμε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν θετικές εξελίξεις το αντίθετο δυστυχώς και βλέπουμε ότι στρέφουμε πολύ λίγο την προσοχή μας σε αυτά τα θέματα και τα υποτιμούμε ή τα υποβαθμίζουμε. Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν για αυτή την κατάσταση. Οι Αμερικανοί δεν έχουν τις καλύτερες επιδόσεις με κανένα τρόπο. Πρέπει συνολικά να δούμε ότι πρόκειται για θέματα ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται, διακυβεύεται έναντι τον ειπα για παράδειγμα που πώς θα αντέξουν οι εταιρείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδου ανταγωνισμό. Και εδώ υπάρχουν πολλά προσκόμματα και εμπόδια. Και σε μια περίοδο κρίση, αυτά τα μέτρα για τα οποία συζητούμε, ακόμα και αν είναι μεμονωμένα μέτρα που άπαξ θα ληφθούν και θα δράσουμε από αυτόν και θα λειτουργήσουν, δεν τηρούμε όμω τι αρχέ για τι οποίε κάνουμε λόγο δίνουμε εξαιρέσεις και κανείς δεν θα μας πιστέψει στο μέλλον ότι με σοβαρό πνεύμα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Οι τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές για το, ε, τον άνθρακα και η ελεύθερη αγορά να τα ρυθμίσει όλα αυτά υπό την λοιπόν, προϋπόθεση κιόλα ότι οι εκπομπές ρήπων είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε σε ακριβότερες ε, κλίμακες να διεξάγεται. Καθίσταται σαφές ότι αυτές οι εκπομπές ρήπων δεν συνδέονται με το καλύτερο τρόπο με τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Στη χώρα μου, στην Πολωνία, έχουμε διαφορετικές, διαφορετικές καταστάσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι τιμέ ενέργειας είναι ένα από τα προβλήματα κλειδιά για μας και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και αυτό θέλω να τονίσω, να προσπαθήσουμε να δούμε, για παράδειγμα, το ότι αυτά τα πιστοποιητικά θα κοστίζουν λιγότερο. Υπάρχει ένας ρόλος ε, που ε, σε σχέση με τα κίνητρα που θα έπρεπε να δοθούν. Υπάρχουν τόσοι πολλοί πολίτες που ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας σε μας ή βρίσκονται πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας είναι πάρα πολύ αρνητική η κατάσταση και πρέπει να διαρωτηθεί κανείς ποια είναι η σημασία όλων αυτών, όχι μόνο για την κοινωνία αλλά και για την βιομηχανία. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο τα χρήματα, τα λεφτά, είναι και μια ιδέα και φυσικά πρέπει να εκφράζουμε και την αλληλεγγύη μας. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε και να μην παίρνουμε στα σοβαρά την αλληλεγγύη. Θέλω να απευθύνω έκκληση οι συνάδελφοι να δουν και βαθύτερα τα αίτια αυτή τη κατάσταση. Έχουμε μία οικουμένη, ένα πλανήτη, όλοι από κοινού και θέλουμε να είμαστε προπομπή στον κόσμο, παγκόσμια. Οι Κινέζοι και οι ΙΠΑ βρίσκονται πολύ πίσω, αλλά πρέπει να λάβουμε πολύ ε, σοβαρά υπόψη τι συμβαίνει γύρω μας για να μην υπάρξουν κάποια παράδοξα. Είναι τέλειο να είμαστε στην Ευρώπη, να έχουμε εκπομπέ ρήπων, που να είμαστε πρωτοπόροι, να είμαστε προπομπή, όμως μας αφήνουν μόνους μας σε αυτή την πορεία οι υπόλοιπε χώρες. Παγκόσμια είμαστε μόνοι μας. Ο Ομπάμα ενδιαφέρθηκε να επανεκλεγεί. Στην Ευρώπη όμως, στην Πολωνία, δεν ε, τηρούνται οι υποσχέσεις που τις δυνατότητες που θα είχαμε θα μας ε, τις ε, ενδυνάμωναν. Ενώ τώρα περιοριζόμαστε και βρισκόμαστε σε ένα πολύ στενό πλαίσιο ε, κινήσεων. Θα πρέπει να δούμε τι είναι δυνατό και εφικτό να γίνει. Να προβληματιστούμε να δούμε. Μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πέτρα λίζες στη συνέχεια. Επόμενος αγορητής. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να θέσω εκ ότι σε αυτό το θέμα δεν παρεμβαίνω ο συντονιστής του ΕΛΚ. Είναι θέμα του Ρίχαρτ Ζέμπερ αυτό. Ήμουν όμως ο εισηγητής της, της Επιτροπής μας για την οδηγία για την αποδοτικότητα στα ενεργειακά θέματα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όλοι από κοινού στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και στην Ολομέλεια ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγίας για την αποδοτικότητα της ενέργειας αλλά και στο πλαίσιο της έκθεσης Chris Davis τον Μάρτιο 2012 εφέτος ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θέματα αυτά να τα εξετάσει και να τα αντιμετωπίσει επιτέλους. Και υπήρχαν και τροπολογίες που ευρύτατα, ευρύτερα υποστηρίχθηκαν. Στο τέλος τέλος στην έκθεση Davis είχαμε συμβιβασμούς μεταξύ ΕΛΚ και ΑΛΔΕ. Αλλά και οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες ενέκριναν την έκθεση αυτή, την υπερψήφισαν. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε. Μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την αποδοτικότητα ενέργεια σε αυτή την οδηγία, έδωσε μια δήλωση, μια διακήρυξη, που πάλι και η Επιτροπή ε, Βιομηχανία και η Ολομέλεια ω μέρο ε, των μέτρων δέσμη ε, τα αντιμετώπισαν. Όποιο μπόρεσε να διαβάσει και να κατανοήσει, τα έλαβε υπόψη αυτά. Σε δύο βήματα, σε δύο φάσει δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό ήταν η εντολή κιόλα. Η εντολή που είχε διαπραγματευτεί σε σχέση με την αντιπροσωπεία μας από διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρώτον, να υποβάλει μια έκθεση για την αγορά άνθρακα, carbon, carbon market και πρόταση για την βελτίωση των πληστηριασμών. Αυτό είναι το backloading. Η ιδέα του backloading είναι κάτι το οποίο από το Κοινοβούλιο προχώρησε και κατανοώ καθέναν που έχει τώρα επιφυλάξεις και λέει ότι είναι λάθος η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατανοώ τα επιχειρήματά τους. Όμως η συζήτηση επί των αρχών, αν θα πρέπει να παρέμβουμε στο σύστημα εμπορία ρήπων ή όχι, έχει διεξαχθεί ω θέμα αρχή σε εμά και στη δική μας Επιτροπή και έχει οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα και σε μία κλίμακα σε δύο βαθμίδες. Πρώτα το backloading και μετά μια συζήτηση που θα διεξαχθεί για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος. Με το backloading εξαγοράζουμε χρόνο και μπορούμε να συζητήσουμε πώς είναι δυνατόν με τον πιο λογικό τρόπο να αρχίσει να μπορέσει να λειτουργήσει με τον πιο συνετό τρόπο το ETS, το σύστημα εμπορίας τρύπων. Είναι καλό αυτό που κάνει ο Ματία. Κάποιε επιφυλάξει και αντιρρήσει σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπής αντιμετωπίζει για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να παρεμβαίνει κάθε εβδομάδα και επανειλημμένα και διαρκώ Και εδώ έχουμε αλλαγή. Άπαξ θα επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πάει πολύ μακριά, διότι δεν μπορούμε προ άλλη κατεύθυνση να αντιδράσουμε. Όμω ίσω αυτό δυστυχώ είναι ανάγκη πλέον να γίνει για να υπάρξει κάποια αποσαφήνιση των όρων του παιχνιδιού Είχαμε συζητήσει πολύ προσεκτικά για το θέμα των διαρροών άνθρακα, carbon leakage, leakage και συζητήσαμε όλα αυτά υπό το πρίσμα μιας μελέτης επιπτώσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να αναμένουμε μια τιμή 30 ευρώ για παράδειγμα για αυτή τη διαρροή άνθρακα, για τα ανθρακικά προϊόντα. Και με την κυρία Κόρολα και εγώ είμαστε κατά της ε, ε, κυρίας Ντόιλ και σε σχέση με το 2008 είπαμε ότι δεν λαμβάνει επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της διαρροής άνθρακα, carbon leakage. Πρέπει όμως να τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Όμως με τιμή 6 ευρώ και όλα αυτά τα οποία αποφασίστηκαν γενικά δημιουργείται πρόβλημα. Και δεν νομίζω ότι ταιριάζουν όλα αυτά και είναι αποτελεσματικά. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά βιομηχανιών, επιχειρήσεων. Είναι δημόσιος ο κατάλογος, έχει δημοσιευθεί μέσα από τη σημερινή κατάσταση έχουμε μια πάρα πολύ ελεύθερη κατανομή και τα benchmarks, οι βέλτιστες αυτές προδιαγραφές θα αρχίσουν να ισχύουν από του χρόνου και έτσι κάποιοι θα έχουν βγάλει εκατομμύρια εκατομμυρίων. Δεν λαμβάνονται λοιπόν επαρκώς κάποια πράγματα από τους σημερινούς κανόνες για το αλουμίνιο για παράδειγμα ή για τον γύψο ε, τα γυψοειδή. Θα πρέπει να πούμε ότι η βιομηχανία μας επιβαρύνεται υπερβολικά λόγω της, ε, του συστήματος εκπομπών, εμπορίας, ε, ε, εμπορίας εκπομπών ρήπων. Το πιο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη σε αυτό το σημείο ξεκινούν να χάνουν ε, τον ρόλο πρωτοπόρου. Εισάγεται ο ρόλος, ε, των, ε, το παιχνίδι των εθνικών τελών και φόρων και αυτό υπονομεύει τα πράγματα. Είναι δηλητήριο. Τα πράγματα αυτά ευρωπαϊκά πρέπει να επιληθούν και όχι εθνικά. Γι' αυτό είμαι υπέρ του να είμαστε μετριοπαθείς, μετριόφρονες, αλλά γοργά να δουλέψουμε. Να μην αναμείνουμε τα κράτη-μέλη εμβαλωματικά να υποβάλουν μια πρόταση συνονθήλευμα εθνικών μέτρων. Έτσι δεν ρυθμίζουμε τα πράγματα. Πρέπει να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, ώστε η αξιοπιστία στην Ευρώπη να αποκατασταθεί και να μην αναλάβουν τα κράτη-μέλη και πάλι τον ρόλο προπομπού. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε εσείς τον λόγο. Είμαι ευγνώμων, λέει ο Λάινεν, στον Πέτερ Λίζε για την παρέμβασή του Πρέπει να υπενθυμίσουμε στη, στην έκθεσή του για την οδηγία αποδοτικότητας ενέργειας όπως και την έκθεση Chris Davis για τον οδικό χάρτη για την ενέργεια μέχρι το 2050 σαφείς τοποθετήσεις γίνονται έγιναν για το σύστημα εκπομπών ρήπων και φοβήθηκα κιόλα σχεδόν από αυτά που άλλοι συνάδελφοι είχαν πει ότι δεν θα κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός αλλά ένα βήμα που θα οπισθοδρομούσαμε προς τα πίσω και αυτό δεν θα ήταν ούτε αξιόπιστο ούτε συνεκτικό και συνεπές. Γι' αυτό ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Πέτερ Λίζε που αφηγήθηκε την ιστορία Πώς δηλαδή την προϊστορία, πώς είδαμε και αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα και πώς στην Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίσαμε και εγκρίναμε κάποια πράγματα. Σύστημα εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα είναι κάτι το καινούριο σχετικά και είναι πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό. Και είναι κάπως, ας το πω έτσι, ένα πείραμα, πειραματικά. Θα δούμε αν λειτουργεί ή όχι και πώς λειτουργεί. Ήδη στο αντίστοιχο άρθρο και στην νομοθεσία είδαμε ότι μπορεί να υπάρχει η αναγκαιότητα, η ανάγκη να υπάρξουν προσαρμογές, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε αυτό το άρθρο 10. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας στον κόσμο. Και η Αυστραλία το εισήγαγε και η Καλιφόρνια και η Νότια Κορέα και μέρος της Κίνας. Και περισσότεροι θα προσθεθούν, διότι η ιδέα ήταν μια παγκοσμιοποιημένη αγορά άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα. Και παρότι ακουγόταν γρίφος αυτό, μπορεί να λειτουργήσει. Και τώρα δεν πρέπει να πετάξουμε τα μέσα και τα εργαλεία αυτά από τα χέρια μας. Πρέπει να γίνουν αποτελεσματικά και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτά. Με 6 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή τη λειτουργία. Λειτουργικά και αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο να υπάρξουν επενδύσεις στις τεχνολογίες και είναι πιο φτηνό να χτίζει κανείς ε, μονάδες που καίνε άνθρακα από το να αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με τις ε, μείωσης των εκπομπών ρήπων. Είναι φθηνότερο να πληρώνει τις εκπομπές ρήπων κανείς δημιουργώντας μονάδες ε, καύσης άνθρακα. Και σε σχέση με τις μελέτες αγορών τι καταδείχθηκε ένα μόνο ευρώ αυξήθηκαν οι τιμές και νομίζω και μειώθηκαν κιόλα εν τω μεταξύ από τότε. Ακόμα και αν εγκρίνουμε τέτοιες προτάσεις το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε, δεν το επιλύουμε. Σε μια δεύτερη βαθμίδα, σε μια δεύτερη κλίμακα θα έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε διαρθρωτικά δομημένα για να τα επιλύσουμε. Πρέπει σε αυτή την έκθεση να παραμείνουμε στα όρια του θέματος και να μην υποβάλουμε τροπολογίες επί του επιστητού για παράδειγμα για αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί σε προηγούμενες ολομέλειες με αποφάσεις μας. Το backloading είναι μια ιδέα, όμως δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όπως δείχνει και η αγορά από τον τρόπο που αντέδρασε δεν αυξήθηκαν οι τιμές. Υπάρχει ένα εγγενές σφάλμα σε αυτό το σύστημα. Όσο περισσότερο εξοικονομούμε ενέργεια, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο λιγότερα τέτοια πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται. Και υπάρχει και πλημμυρίδα τέτοιων πιστοποιητικών στην οποία καταλήξαμε. Έχουμε υπερβολικά πολλά τέτοια πιστοποιητικά και πρέπει κάποιες άλλες σκέψεις να κάνουμε για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ε, ε, έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Και τώρα θυμάμαι κάτι άλλο. Όχι μόνο τα πιστοποιητικά αυτά αφορούσαν τις ίδιες τις βιομηχανίες που ήταν ηρυπαίνουσες, αλλά είχαμε ολόκληρη αγορά οικονομική με τέτοια πιστοποιητικά. Ανοίγει πόρτα εδώ για κάθε είδους παρατυπία και απάτη. Κλέβουν κάποιοι κάποια τέτοια πιστοποιητικά. Ελπίζουμε να γίνει πιο στεγανό αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν κάποια διπλά πιστοποιητικά που κυκλοφορούν στην αγορά. Φοροαπάτη διεξάγεται με τέτοιου είδους κυρίως η Deutsche Bank κιόλα, σε μια ε, επιδρομή που έγινε από την αστυνομία, ε, διαπιστώθηκε ότι είχε συμμετάσχει σε τέτοιες απάτες κατά πολύ μεγάλο όγκο χρημάτων, 230 εκατομμύρια λέει ο μιλητής και ποτέ δεν πρόκειται σε σχέση με την Barclays Bank να αναφερθούμε σε ε, δική της τοποθέτηση. Πρόκειται για τράπεζα καζίνο. Δεν είναι εδώ για προστασία του περιβάλλοντος αλλά για κερδοσκοπία και μάλιστα με σχροκέρδια με την οποία κινούνται. Μόνο το κέρδος τους ενδιαφέρει από ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Πώς μπορούν να πετύχουν κάποια δισεκατομμύρια κέρδους. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί έναντι των κόλπων που κάνουν η τράπεζα Μπάχλης και άλλοι. Παρ' όλα αυτά λοιπόν το πρόβλημα υπάρχει, υφίσταται με αυτή την έκθεση νομίζω κάνουμε ένα πολύ μικρό βήμα. Ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, άλλα βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οπωσδήποτε. Ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης επόμενος, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση που έχω. Άκουσα ότι είναι πολύ καλό να έχουμε υψηλές τιμές σε αυτή την αγορά. Και αναρωτιέμαι οι προσπάθειές μας ε, αποσκοπούν σε υψηλές τιμές ή προς μια αγορά που να λειτουργεί σωστά και να αποδίδει όπως πρέπει. Έχουμε ύφεση. Ήφεση σημαίνει ότι οι τιμές πέφτουν και έχουμε και το σκάνδαλο CDM που επίσης βοήθησε να χαμηλώσουν οι τιμέ. Αλλά το ότι οι τιμές χαμηλώνουν δεν σημαίνει ότι δεν, δεν, σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους. Σημαίνει ότι επιτυγχάνουμε υπερβολικά τους στόχους. Όχι γιατί το θέλαμε, αλλά γιατί έτσι συνέβη. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν σήμερα ανεβάσουμε τις τιμές θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις. Αλλά αυτό που προτείνεται είναι να ανεβάσουμε σήμερα την τιμή και να τη χαμηλώσουμε το 2019 και το 2020. Και η ερώτηση είναι, εάν μιλάμε για μελλοντικές επενδύσεις, και υποθέτω ότι γι' αυτό μιλάμε, γιατί πιστεύουμε ότι το να χαμηλώσουμε την τιμή το 2020 θα βελτιώσει τις επενδύσεις. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Τότε θα ξεκινήσουν να αποδίδουν οι σημερινές επενδυτικές αποφάσεις οι σημερινές επενδυτικές αποφάσεις δεν έχουν σχέση με το τι θα συμβεί στα επόμενα τρία χρόνια. Μια επενδυτική απόφαση σήμερα θα αρχίσει να αποδίδει μετά από πέντε χρόνια. Σε χαμηλότερη τιμή δηλαδή. Για ποιο λόγο λοιπόν συμβαίνει αυτό. Μήπως γιατί ορισμένες χώρες ε, θέλουν να παρέχουν κρατική ενίσχυση στην και τους βιομηχανία. Μήπως διότι κάποιες άλλες χώρες θέλουν να φορολογήσουν και να ρίξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, το πολιτικό κόστος, διότι μιλάμε για πολλά λεφτά. Το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο δημοσίευσε μια εκτίμηση. Μια εκτίμηση για το κλίμα και την ενέργεια από το αντίστοιχο τμήμα, όπου αναφέρεται ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση αν δεν κάνουμε απόσυρση από φόρων. Στη χώρα μου, εάν δεν κάνουμε αν αποσύρουμε 900 εκατομμύρια τόνους μαζί με το 2020 θα ε, μιλάμε για ποσό 3,3 δις. Μιλάμε για πολλά λεφτά όσον αφορά τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος ε, και άλλες χώρες θα έχουν δυσκολίες. Θα πληρώσουν πολλά λεφτά αν αυτό συμβεί. Σύμφωνα με το Ρωμανό οι χώρες οι οποίες θα πληρώσουν περισσότερο θα είναι η Ρουμανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Ισπανία. Οι φτωχοί της Ευρώπης θα πληρώσουν πολλά λεφτά σε λογαριασμούς ηλεκτρικού. Για ποιο λόγο. Και η Γερμανία επίσης. 19 δις λέει το Ηνωμένο Βασίλειο εάν εάν βγάλουμε 900 εκατομμύρια τόνου ανεπιστρεπτή. Δεν ξέρω αν αυτέ οι εκτιμήσει είναι σωστέ, μπορεί να είναι και λάθο οι αγορέ, είναι δύσκολο να προβλεφθούν, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι πολίτε μα θα πληρώσουν το κόστο των αποφάσεών μα. Ένα τεράστιο νέο φόρο. Γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν θα επηρεάσει τι μελλοντικέ επενδύσει, θα επηρεάσει τι επενδύσει των επόμενων δύο ετών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, τα πιστοποιητικά αυτοκίνητα αυτόματα σε σχέση με τις τιμές που καταβλήθηκαν, αυτόματα λειτουργήσαν. Αυτό είναι το μάθημα το οποίο μάθαμε από την πρώτη περίοδο εμπορίας, ότι είχαν δοθεί δωρεάν αυτά, όμως οι επιχειρήσεις ε, καθόρισαν τιμές. Ε, ήδη πλήρωσαν λοιπόν έτσι οι καταναλωτές. Κορίν Λεπάζ παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα, διότι πολύ συγκεκριμένα το σύστημα που έχουμε υλοποιήσει δεν μας επέτρεψε να επιτύχουμε τους στόχους που θέλαμε. Πολύ απλά διότι ήμασταν υπερβολικά ελαστικοί όσον αφορά τον αριθμό πιστοποιητικών που εκχωρήσαμε, ποσοστόσων που εκχωρήσαμε στις βιομηχανίες. Δηλαδή τα κράτη και κυρίως το δικό μου κράτος, όπως είδα, παρήχαν ποσοστώσεις ε, που είχαν προβληθεί για τις επιχειρήσεις πολλές περισσότερες από τις απαραίτητες για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη και ξαφνικά βρισκόμαστε με πλεόνασμα προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση με αποτέλεσμα να καταρακώνονται οι τιμές. Πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε σε έναν οικονομικό ρεαλισμό αυτό των ποσοστώσεων που έπρεπε να κατανεμηθούν φυσιολογικά όπως πολλοί συνάδελφοι και εγώ ε, με απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της βιομηχανίας μας και της ανταγωνιστικότητάς της στη βιομηχανία. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλοί βιομηχανικοί τομείς. Για να έχουμε συνοχή με αυτά που λέμε και με τις ε, πολιτικές που θέλουμε να διεξάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά το 3 επί 20, είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές τιμές ε, ενώπιον των νέων βιομηχανιών που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να, αναπτυχθεί, να αναπτυχθούν αυτοί οι τομείς αποδοτικά θα πρέπει η τιμή του άνθρακα να αντιστοιχεί σε κάτι. Αλλιώς ε, δεν θα αποδώσουν. Το είπα και προηγουμένως. Ε, το είπαμε και προηγουμένως. Είναι ε, πιο φθηνό να κάνουμε θερμικές βιομηχανίες άνθρακα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι παράλογο. Συνεπώς, ε, εγώ υποστηρίζω αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ρωτάω είναι μέχρι πού πρέπει να το πάμε. Ε, έχουμε δει διάφορες αξιολογήσεις αντικρουόμενες όσον αφορά το τι χρειάζεται. Άλλες φορές μας λένε 900.000, την άλλη φορά μας λένε 1 δις 8. Ε, εγώ δεν ξέρω ακριβώς τι να σκεφτώ. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συζητήσουμε πριν συμφωνήσει η Επιτροπολογία παρά να συζητάμε επί της αρχής. Η αρχή είναι ε, προφανής. Να δούμε πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον των ε, ευρωπαϊκών βιομηχανιών που θέλουν να διεισδύσουν σε αυτές τις νέες αγορές ή να είναι ηγέτες αυτών των νέων αγορών. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο σε αυτή την αρχή του 21ου αιώνα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η Φρανσουάς Γκροστέτ παρακαλώ έχει τον λόγο. Merci, merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μελετώντας την έκθεσή σας, παρατηρούμε ότι η θέση σας ε, είναι σοφή, διότι προτείνεται να καταφύγουμε σε μία μόνο προσαρμογή της Κομισιόν για την περίοδο 2013-2020 για τους πληστηριασμούς. Ε, φαίνεται ή να είναι μέσα σε άκρηση ικανοποιητική αυτή η πρόταση, σε άκρη ικανοποιητικη επιτρέπει προβλεψιμότητα για τις βιομηχανίες. Παρατηρώ ωστόσο ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μπορεί να παρέμβει ανα πάσα στιγμή όσον αφορά την απόσυρση ποσοστώσεων χωρίς καθαρή εντολή, ε, καταφεύγοντας τον backloading. Μελετώντας κάπως τα πράγματα, ανησυχώ παρόλα αυτά. Ανησυχώ διότι Φυσικά αφενός μιλάμε για το τεράστιο πλεόνασμα ποσοστώσεων που οδηγεί σε μείωση των τιμών του άνθρακα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Φυσικά παρόλα αυτά διερχόμαστε μια περίοδο βαθιάς κρίσης. Αυτή η κρίση αιτιολογεί τη μείωση των τιμών του άνθρακα. Είχαμε πολύ χαμηλότερου ρήπου από ό,τι φανταζόμασταν. Και φυσικά η αγορά όπως είχε δημιουργηθεί, όπως σχηματίστηκε, όπως διαμορφώθηκε, οδήγησε σε αυτή τη μείωση το τιμό του άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ήθελε να προτείνει ένα σύστημα βασισμένο στη λογική της αγοράς και σήμερα λέει ε, λοιπόν εγώ θα το ρυθμίσω. Θα το ρυθμίσω και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την ελευθερία να προβεί σε παρεμβατισμό. Δηλαδή μια απολύτω ελεύθερη κομισιόν ξαφνικά θέλει να παρέμβει. Εμένα με ανισχύει αυτό διότι οι βιομηχανίες χρειάζονται σταθερότητα, ειδικότερα αυτή την εποχή τη ύφεση. Πιστεύω λοιπόν ότι λογικό θα ήταν να διατηρήσουμε τους τρέχοντες κανόνες μέχρι για την περίοδο 2013-2020 ώστε να διατηρήσουμε αυτή τη νομική βεβαιότητα, σταθερότητα για τους ενδιαφερόμενους. Διότι ούτως ή άλλως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης με αυτό το σύστημα, για αυτό το σύστημα ETS. Πιστεύω ότι το να αρχίσουμε να αμφισβητούμε όλα αυτά σήμερα στο τρέχον πλαίσιο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αρνητική αντίληψη, σε μια αρνητική αντιμετώπιση από τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις. Ας προσέξουμε λοιπόν, η θέση της Κομισιόν δεν με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάισκεμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν, Πρόεδρε, το βρίσκω πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για το μέλλον του συστήματος εμπορίας τρύπων και να προβληματιστούμε σε βάθος τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να διασφαλίσουμε, θα έλεγα, ότι αυτό το σύστημα θα παραμείνει και θα μπορέσει να λειτουργεί αποτελεσματικά και στο μέλλον. Και γι' αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό, μόνο σημαντικό να έχουμε οικονομικά κίνητρα για καινοτομία και δράση, αλλά και για την πλευρά των εσόδων από το ETS, από την εμπορία ρήπων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατεπηγόντως αυτά τα έσοδα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών για να έρθουμε στη σωστή πορεία. Και μπορεί κανείς ήδη κιόλα να διαπιστώσει και να πει ότι οι χαμηλές τιμές που ισχύουν σήμερα <clears throat> για δικαιώματα ρήπανσης που πληρώνονται σήμερα δεν ανταποκρίνονται και δεν δικαιώνουν αυτούς τους δύο στόχους που θα έπρεπε να λειτουργήσουν καλύτερα. Από πλευράς αρχής λοιπόν η ιδέα του backloading μπορεί να υποστηριχθεί και αξίζει να υποστηριχθεί. Υιοθετώ όμως μια μεσαία θέση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων για την μία που απορρίπτουν και για τους άλλους που είναι απλά υπέρμαχοι. Νομίζω ότι και ο εισηγητής βρίσκεται στη μεσαία αυτή γραμμή πλεύσης και θα ήθελα αυτό να το αναγνωρίσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία με αυτή την προσέγγιση. Πρώτον, δεν μπορεί να, να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καταφέραμε αυτό εμείς. Δεύτερον, είναι σημαντικό όχι μόνο μια προσαρμογή να έχουμε σε σχέση με το 2013-2020, προσαρμογές δηλαδή που θα είναι εφικτές σε σχέση με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αποσαφήνισε αυτό ο εισηγητής. Πρέπει να μιλήσουμε και για άλλους όρους και προϋποθέσεις πιστεύω, που σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε εδώ ότι δημιουργούν ένα πλαίσιο που περιορίζουν τις κινήσεις ε, στην ε, αγορά όσον αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν. Θέλαμε να, είχαμε, να έχουμε ένα μέσο διαχείρισης και αντιμετώπισης. Ερωτώ τον εισηγητή, θα μπορούσε να εξετάσει ενδεχόμενα την δυνατότητα μιας επαναγοράς αν για παράδειγμα υπάρχει ξαφνική άνοδος ή ξαφνική αλλαγή των τιμών, ε, μεταβολή των τιμών, θα ήθελα να ακούσω την άποψή του. Δηλαδή, ήδη προβλέπεται κάποια τέτοια κίνηση στην έκθεσή του ή σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπόρεσα να το συναγάγω εγώ αυτό. Τι θα μπορούσε να γίνει και πώ δηλαδή μέσω άλλων όρων και προποθέσεων που θα προσαρμόζαμε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για αυτή την παρέμβαση ή επέμβαση, γιατί για επέμβαση πρόκειται, που να κρατούσαμε αυτή την επέμβαση στο δυνατόν στενότερο και πιο ε, καθορισμένο, περιορισμένο πλαίσιο. Και κάτι άλλο, επιτρέψτε Πρόεδρε, που είναι σημαντικό για μένα. Μέσα σε αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συζητήσουμε ένα πράγμα. Το ανέφερε και ο συνάδελφος ότι ο μηχανισμός διαρροής άνθρακα είναι άδικος. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες εξαιρέσεων που έχουν κάποιο νόημα και μπορεί να είναι ε, δίκαιοι. Όμως εξαιρούνται κάποιοι βιομηχανικοί κύκλοι που βρίσκονται σε στενό ανταγωνισμό με άλλους βιομηχανικούς κύκλους και δραστηριότητες που δεν εξαιρούνται και που μάλλον κιόλα παράγουν προϊόντα τα οποία βρίσκονται ανταγωνιστικά στην αγορά έναντι άλλων προϊόντων και, έχουν, και ευνοούνται κιόλα. Κάτι τέτοιο δεν θα είχε κανένα νόημα να γίνεται. Για παράδειγμα, σε σχέση με τον ε, τομέα των ε, γυψικών προϊόντων και εδώ θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Δεν θέλω να ασκήσω κάποιε επικρίσεις, αλλά τα προϊόντα να τα συγκρίνουμε, όταν τα συγκρίνουμε βλέπουμε ότι είναι πιο αποτελεσματικά αποδοτικά σε σχέση με την χρήση ενέργειας α, τέτοιου είδους προϊόντα. Πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις λοιπόν. Καλό θα ήταν αν μια τέτοια θέση επί της αρχής προβλέπαμε από πλευράς έκθεσης. Αν ήσουν ανοιχτός εσύ εισηγητή για κάτι τέτοιο, αυτό το μηχανισμό carbon leakage, διαρροή άνθρακα, θα έπρεπε να το καταστήσουμε πιο δίκαιο και πιο σωστό για το περιβάλλον, να μην υπάρχουν αδικίες δηλαδή σε σχέση με αυτόν. Ευχαριστώ Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Chris Davis, τελευταίος αλλά σημαντικός πολύ. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα κύριε Πρόεδρε, πέρασα από την Επιτροπή Αλίας ε, για κάποιες ψηφοφορίες που θα γίνουν αύριο έπρεπε να βρίσκομαι εκεί. Λοιπόν, έχασα ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης, αλλά γνωρίζω ότι πολλοί συζήτησαν για την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτή την νομοθεσία πολύ απλή νομοθεσία για να αναθεωρήσουμε ολόκληρο το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών και να προσθέσουμε την απέτηση παρακολούθησης από την Κομισιόν κάνοντας προτάσεις ε, για να βγάλει δικαιώματα από την αγορά και όλα αυτά. Εγώ απορρίπτω όλες αυτές τις ιδέες. Εγώ είμαι τη άποψη ότι αυτή η πρόταση είναι απλή και πρέπει να διατηρηθεί απλή. Έχουμε τον οδικό χάρτη για τι χαμηλέ εκπομπέ ρήπων. Το έχουμε δηλώσει σαφώ και σε αυτή την επιτροπή και στην επιτροπή Ίντρα. Ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πράγματα πιο πολύπλοκα και να το κάνουμε μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα από ό,τι πρέπει να είναι. Λέγεται ότι δεν πρέπει να δώσουμε λευκή κάρτα στην Κομισιόν. Αλλά το γεγονός είναι ότι η Κομισιόν έχει στραφεί προς εμάς με αποφάσεις ε, συναπόφασης ουσιαστικά, με νομοθεσία συναπόφασης. Ε, αυτό το χρονοδιάγραμμα για τα δικαιώματα δεν αλλάζει ο ρυθμός των δικαιωμάτων ουσιαστικά που θα υπάρχουν στην αγορά. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Κομισιόν είναι ρυθμιστική αρχή. Είναι κάτι σαν ρυθμιστική αρχή και πρέπει να της επιτρέψουμε να κάνει τη δουλειά της όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του ETS θα τα συζητήσουμε αργότερα, του χρόνου. Και αναμένω η Κομισιόν να κάνει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, εμπορίας εκπομπών, έχει αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Έχουν μειωθεί οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Ίσως να ζητάμε υπερβολικά πολλά όταν υποθέτουμε ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να παρέχει επίσης και επενδύσεις ε, σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Πρακτικά δεν έγινε αυτό έτσι. Επιτευχθεί μέσω ρυθμίσεων για, τα, ε, για τους υδροχλωροφθοράνθρακες, για παράδειγμα, με τον ορισμό συγκεκριμένων στόχων. Αλλά πολύ λίγα ε, μπορούν να αποδίδονται στο ETS άμεσα. Να μην το αναμένουμε αυτό δηλαδή για το μέλλον. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, πιστεύω, είναι ότι αναγνωρίζουμε ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι το βασικό μέσο της Ευρώπης για την καταπολέμηση ε, των αερίων θερμοκηπίου από τις βιομηχανίες. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλές άλλες χώρες ολόκληρο τον κόσμο σήμερα προσπαθούν να αντιγράψουν το δικό μας μοντέλο. Θα ήταν λάθος να αφήσουμε να καταρρεύσει το ETS. Αυτό είναι ο κίνδυνος ο κίνδυνο είναι ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί στι αλλαγέ ε, που θα επιφέρει το backloading και αν εμεί ε, ε, εναντιωθούμε σε αυτέ τι προτάσει, τότε η εμπιστοσύνη στο σύστημα αυτό θα καταρρεύσει σχεδόν ολοκληρωτικά. Η επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, μου είπε, ένας εκπρόσωπός μου είπε προσωπικά πριν από μερικούς μήνες πραγματικά δεν μας αρέσουν αυτές οι προτάσεις backloading αλλά μας αρέσει η ιδέα του να μην υπάρχουν αυτές οι προτάσεις αλλά η ιδέα του να μην υπάρχουν αυτές οι προτάσεις δεν μας αρέσει ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, ας διατηρήσουμε λοιπόν για να έχουμε περιθώριο δράσης. Ευχαριστώ και για αυτή την καταληκτική παρατήρηση και δίνω τον λόγο στην επικεφαλής μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή αυτών των ιδεών. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από πλευρά μα. Φυσικά διαβάσαμε προσεκτικά την έκθεσή σα. Θα ήθελα απλά να υπενθυμίσω κάποια σημεία που υποστηρίζουν την πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση του ε, χρονοδιαγράμματος πληστηριασμών η Κομισιόν ε, πάντα εξέφρασε ότι δεν είχε ιδιαίτερη προτίμηση προς αυτή την πρόταση. Χρειάστηκε λίγο χρόνο. Κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση για backloading 900.000 δικαιωμάτων αλλά η συζήτηση ε, ε, ε, αναφέρθηκε σε συνδέσεις μεταξύ του ETS και άλλης νομοθεσίας ε, όταν προτάθηκε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πακέτο για την ενέργεια. Υπήρξαν αυτές οι διασυνδέσεις ε, ενσωματωμένες σε αυτή την πρόταση. Τώρα το θέμα είναι οι προτάσεις για την ενεργειακή απόδοση. Εκεί πολλά μέλη του παροντό κοινοβουλίου υπενθύμησαν τις διαπραγματεύσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και τη κατεύθυνση που δόθηκε εκείνη τη στιγμή όταν η Κομισιόν δεσμεύτηκε για την έκθεση και κοίταξε για αναθεώρηση των πληστηριασμών. Αυτό ακριβώς κάναμε και γι' αυτό το λόγο επιμένουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη σημαντική κατάσταση. Το πλεόνασμα το οποίο εμφανίστηκε επίσης λόγω και άλλων ρυθμιστικών αποφάσεων που λήφθηκαν μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζω και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όλοι μαζί αποφασίσαμε να περιορίσουμε τον αριθμό πιστώσεων στο μηχανισμό καθαρή ανάπτυξη που θα χρησιμοποιηθεί στο ETS και κυρίω όσον αφορά του υδροχλωροφθοράνθρακες. Όπω ξανά έχει ξανααναφερθεί αυτέ οι αποφάσει. λένε ότι οι πιστώσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμμόρφωση μόνο για το 2012 το αργότερα και όλε αυτέ οι πιστώσει θα χρησιμοποιηθούν και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αντίστοιχο πλεόνασμα δικαιωμάτων εφόσον οι πιστώσει και τα δικαιώματα προστίθενται, αθρίζονται πέραν αυτών ε, έχουμε και την οικονομική κρίση όπως αναφέρατε πολλοί από εσά και αυτό είναι κάτι που απλά πρέπει να δεχτούμε ότι δεν το είχαμε προβλέψει όταν συμφωνήσαμε το πακέτο κλίματος και ενέργειας και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να αυτό, διασφαλίζει αυτή τη συμφωνία. Ε, εδώ μιλάμε για ένα προσωρινό μέτρο, το υπενθυμίζω. Η Κομισιόν ταυτόχρονα έχει κάνει την έκθεση για περισσότερα δομικά μέτρα, ενίσχυση του ΙΤΕΣ e και εμεί χαρούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και το 2013. Στο μεταξύ, έχουμε ξεκινήσει διαβούλευση με του ενδιαφερόμενου για αυτή την έκθεση, ώστε να συζητήσουμε τι επιλογέ και θα οργανώσουμε επίση και μια σειρά από συνεδριάσει με ενδιαφερόμενου. Απλά να υπενθυμίσω γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την ε, αναθεώρηση των πληστηριασμών πρώτα απ' όλα για να επαναλάβουμε τα όσα είπατε πολλοί από εσά. Δεν είναι βέβαιο πώ θα επηρεαστούν οι τιμέ του άνθρακα από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε στην εκτίμηση αντικτύπου μα για την πρόταση backloading ε, παρέχει κάποια αποτελέσματα που μας πρότειναν οι αναλυτέ αγοράς. Κάποια εύρη τιμών. Αναμένεται λοιπόν ότι η επιρροή δεν θα είναι πολύ μεγάλη και σίγουρα κάτω από το εύρο που σκεφτόντουσαν ο καθένα και που συζητήθηκαν στι διαπραγματεύσει για το πακέτο, για το κλίμα και την ενέργεια. Από την άλλη, άλλοι αναλυτέ αγορά λένε ότι η τρέχουσα τιμή του 6,55 ευρώ ήδη λαμβάνει υπόψη αυτή την έννοια του backloading και ότι αν αυτή η πρόταση δεν εγκριθεί οι τιμές μπορεί να πέσουν και άλλο. Και αυτό πιστεύω είναι άλλο ένα επιχείρημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, όπως είπατε πολύ, και πιστεύω αυτό αποτελεί την κύρια αιτία για την πρόταση της Επιτροπής, είναι το να διατηρήσουμε τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Έχουμε όλοι συζητήσει εδώ και πολύ καιρό τον οδικό χάρτη χαμηλών εκπομπών άνθρακα για στον ορίζοντα 2050 Συζητήσατε μόλι και τα αποτελέσματα τη Ντόχα και ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε φιλοδοξίε. Πιστεύω είναι σημαντικό να διατηρούμε στο νου μα ότι αν συνεχίσουμε με τι σημερινέ τιμέ, αυτό θα εμποδίσει τι επενδύσει σε οικονομία χαμηλών εκπομπών που όλοι χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το διατηρούμε στο νου μα και αυτό μα λένε και ενδιαφερόμενοι. Ότι η τιμή αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι αναμενόταν. Αυτό είναι φυσιολογικό σε κάποιο βαθμό τη οικονομικής κρίσης, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω και θα πρέπει να λάβουμε μια λογική απόφαση το να διευρύνουμε το ποσό των δικαιωμάτων ε, περισσότερο, με λογικό τρόπο. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι η επιρροή στα έσοδα. Αυτά τα δικαιώματα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των κρατών μελών και όταν τα βάζουμε στην αγορά με τέτοιε τιμέ, αυτό θα επηρεάσει και τον προπολογισμό των κρατών μελών και το πώ είχαν προγραμματίσει να ε, χρησιμοποιήσουν αυτά τα έσοδα για να προωθήσουν τι κλιματικέ επενδύσει και τι επενδύσει σε ενεργειακή απόδοση. Ένα άλλο σημείο που αναφέρθηκε, το οποίο παρατηρούμε και εμεί αυτή τη στιγμή, είναι ότι αν οι τιμέ παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται και το backloading δεν υλοποιηθεί, τότε πράγματι, και αυτό συμβαίνει ήδη σε ορισμένα κρατημέλη, θα υπάρξουν πρόσθετα εθνικά μέτρα και εσεί το αναφέρατε κύριε Λίζερ, θα υπάρξει κατακαιρματισμό τη εσωτερική αγορά με αρνητικέ επιπτώσει σε όσου συμμετέχουν στο ETS. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω, θέλω να σας τονίσω ότι σε σχέση με τις τροπολογίες σας, ειδικότερα την 6 και την 4, έχουμε κάποιους ενδιασμούς. Θα επαναλάβω ότι η Κομισιόν έχει αφοσιωθεί πλήρως στην αναθεώρηση του προφίλ ε, ε, για τα auction, για του πληστηριασμού μόνο σε εξαιρετικέ περιπτώσει και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εξαιρετικέ περιπτώσει. Πριν από τέσσερα χρόνια, όπω είπα, κανεί δεν θα μπορούσε να έχει φανταστεί την σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό το να περιορίσουμε την κατεξουσιοδότηση, της κατεξουσιοδότηση πράξη σε μόνο μία φορά θεωρούμε ότι δημιουργεί πρόβλημα στην αναθεώρηση των πληστηριασμών, του προφίλ πληστηριασμών, πάντα θα εμπλέκεται η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Και μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι μιλάμε για εξαιρετικέ περιστάσει, μόνο σε τέτοια περιπτώσει θα μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια αναθεώρηση. Για ολόκληρη τώρα τη φάση 3 να αναθεωρήσουμε αυτό το προφίλ πληστηριασμών πιστεύουμε ότι είναι λίγο προβληματικά. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν μετά από συζητήσει με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε επίσημες θέσεις. Και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Φυσικά μπορώ να κατανοήσω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τις δύο τροπολογίες αυτές, την 4 και την 6, δεν, μπορώ, δεν τις θεωρείτε, δεν τις αντιμετωπίζετε με θετικό πνεύμα. Όμως ενέταξα όλα αυτά που στην πρώτη συζήτηση απέρευσαν και παρουσιάστηκαν ως επιχειρήματα. Θεώρησα ότι ήταν σημαντικό, μια και πρόκειται για μια άπαξ δράση, να υπάρξει μετά στη συνέχεια ανυφαλιότητα και ηρεμία και να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν που συσχετίζονται όχι αρχικά ως ε, ζητήματα με αυτή την έκθεση, αλλά αναφέρονται και τα θέματα των ε, επιχειρήσεων εντατικής εκμετάλλευσης και καταδείχθηκε σαφώς ε, και με την έκτακτη συνεδρίαση που είχαμε ως Επιτροπή, όπως αποσαφηνίστηκε σαφώς ότι ο κατάλογος των εντατικών αυτών επιχειρήσεων και ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κατάλογος. Κάποιοι δεν συμπεριλαμβάνονται εκεί που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται. Έχουμε όμως και ε, διάφορες παραγωγές. Ε, εταιρείε, ε, διάφορες εταιρείε που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ίσως σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσουμε. Και οι συντονιστές αποφάσισαν τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο την έκθεση για το διοξίδιο του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τη συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με την Ιρλανδική Προεδρία. Να δώσουμε προσανατολισμούς. Τι θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον με την αγορά διοξιδίου του άνθρακα και άνθρακα ως Ευρωκοινοβούλιο. Το επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή θέση εδώ να τα εντάξουμε όλα αυτά. Να μην υπερβαρύνουμε αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά και στην Ολομέλεια. Χρειάζεται προσανατολισμού η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ καλούνται οι συντονιστέ να δράσουν. Πώ δηλαδή θέλουμε να λειτουργήσει αυτή η ε, δράση από πλευρά μα. Οι εξαιρέσει είναι υπερβολικά ευρείε και κάποιοι που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται δεν συμπεριλαμβάνονται. Έγιναν σφάλματα λοιπόν και πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικές δράσεις για βελτιώσεις. Εδώ αλληλεγγύη αναφέρθηκε ως όρος. Θα ήθελα να πω να προσέξουμε. Αν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε την Ευρω... τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, να ανακάμψουν και σε όλους τους τομείς πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, να υπάρξουν προσαρμογές, συντονιστικό έργο. Η αγορά του διοξιδίου του άνθρακα, του άνθρακα πρέπει να βελτιωθεί, να ρυθμιστεί καλύτερα. Είχαμε μια κρίση που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Και όλα αυτά κανένας δεν τα είχε προβλέψει όταν εμείς ε, καθορίζαμε και εκπονούσαμε τους κανόνες και κανονισμούς ως κοινοβούλιο, υπερβολικά εξειδικευμένα ως κοινοβούλιο, αλλά αποσαφηνίστηκε αυτό και το είδαμε όταν με τους ε, Κινέζους συναδέλφους συζητήσαμε αυτά τα θέματα. Είδαμε ότι σε επτά περιφέρειες ε, ξεκινούν με ένα τέτοιο σύστημα εμπορίας ρήπων και θα έχουμε και ένα σύστημα κινέζικο εμπορίας ρήπων που θα προχωρήσει. Ας αναμείνουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ήταν ανοιχτοί οι Κινέζοι να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους σε αυτό το πεδίο και η προστασία για το περιβάλλον μόνο παγκόσμια μπορεί να λειτουργήσει. Και αν έχουμε παρόμοιες και όμοιες προϋποθέσεις και ρυθμίσεις, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά. Μόνο με το σύστημα εμπορίας ρήπων μπορούμε να προχωρήσουμε. Εύχομαι περαστικά και καλή επιτυχία σε όσους θέλουν να εισαγάγουν ένα τέλος διοξιδίου του άνθρακα. Δεν το καταφέρνουμε ούτε στην ε, Ευρωομάδα ή στην ε, ομάδα των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι τέτοιο να το προχωρήσουμε γοργά. Και γι' αυτό παρακαλώ παρακαλώ θερμά αυτά τα οποία από κοινού επί χρόνια ρυθμίσαμε και αποφασίσαμε για να ε, υπάρξει ρύθμιση της αγοράς ε, πρόθεσμα να διεξαγάγουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μια συζήτηση, να ξεκινήσουμε στις αρχές του χρόνου, το 2013, όχι εδώ, σε αυτό το σημείο, υστερότερα θα συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει, ώστε αυτή η αγορά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να ρυθμιστεί και να λειτουργεί καλά. Και Αναφέρθηκε και από συναδέλφους σε αυτό το θέμα. Ανώτερες και κατώτερες οροφές, ε, ανώτερα όρια, κατώτερα όρια. Θα μπορούσα να φανταστώ, όχι σε αυτή την έκθεση, αλλά αλλού, να το συζητήσουμε αυτό να έχουμε για παράδειγμα όπως και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα διοικητικό συμβούλιο, ένα συμβούλιο όπως και η Αυστραλία για παράδειγμα θα ενταχθεί ή θα θέλει να συμμετάσχει να υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο θα συζητά και θα βλέπει πώς θα είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις και θα θέτει ανώτερα κατόφλια και κατώτερα ανώτερα ανώφλια και κατώτερα κατόφλια ως οριακές τιμές. Καλό θα ήταν να έχουμε έτσι αυτό, ε, ένα πλαίσιο ε, που θα ρυθμίζαμε για αυτές τις ε, δραστηριότητες. Να έχουμε ένα ισοδίκιο πεδίο δράσης και σαφείς κανόνες και κανονισμούς. Προς όλους εκείνους που έχουν αμφιβολίες κατέστη σαφές από συναδέφους, εμείς εμείς ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Δεν το έκανε εκείνη ε, θελούσια και επειδή έτσι έτυχε. Εμείς επανειλημμένα διάφορες φορές και σε διάφορα νομοθετικά πεδία με διάφορες διαφορετικές εκθέσεις ζητήσαμε πλειοψηφικά να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκανε τη δουλειά της πριν από τις θερινές διακοπές. Και εγώ από τους συντονιστέ έλαβα την εντολή αυτή την έκθεση να την συντάξω με τροπολογίε. Υπήρξε συζήτηση αν θα έπρεπε να συντάξουμε τροπολογίε ή όχι. Είπαμε πλειοψηφικά ότι θέλουμε να ενταχθούν όλα αυτά σε μια λογική διαδικασία κοινοβουλευτική για να τα ρυθμίσουμε. Αυτό κάνουμε. Προσβλέπω να δω ποιε θα είναι οι λίγε τροπολογίε αυτέ που θα κατατεθούν και απευθύνω έκκληση στο τέλο ομοιοπαθητικέ δόσεις ε, να ε, έχει αυτό το φάρμακο, αυτή η πρόταση, ώστε να καταλήξουμε σε μια λογική συμβαστική λύση, σε ένα συμβιβασμό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το backloading. Και μετά ύστερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με άλλε προτάσει όπου θα συζητηθούν στην Επιτροπή μα και θα δούμε πόσα πιστοποιητικά θα αποσυρθούν από την αγορά στο τέλος τέλος. Και τρίτον, η έκθεση για την αγορά άνθρακα που αναφέρεται και με τις έξι εναλλακτικέ προτάσεις ή λύσεις. Να δούμε, μήπως θα πρέπει να προσθεθούν και άλλες εναλλακτικέ δυνατότητες εδώ. Και ζήτησε κάποιος συνάδελφος, κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν να παρέμβουν. Καλό τους συναδέλφους αυτούς στην Ολομέλεια να παρέμβουν. Όταν θα έχουμε αυτή την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και επικοδομητικά να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά γενικά, αυτά που ήθελα να πω για αυτό το θέμα. Και καταληκτικά ολοκληρώνω προ το Συμβούλιο, δεν ξέρω, υπάρχει εκπρόσωπο του Συμβουλίου, να πείτε στου συναδέλφου στο Συμβούλιο ότι αναμένουμε από το Συμβούλιο να σημειωθούν πρόοδοι και ιδιαίτερα από τη δική μου χώρα, κράτο μέλο, τη Γερμανία. Υπάρχει εκεί αντιπαράθεση. Έχουμε παράδοση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντο και Υπουργείου Βιομηχανία. Δεν έχει μια τέτοια συντονισμένη θέση η Γερμανία. Και ω μεγαλύτερη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συντονιστεί, να έχει μια λογική λογική ρυθμισμένη η τέτοια πρόταση ώστε αυτό το backloading να μπορέσει να λειτουργήσει και όλα τα υπόλοιπα μέτρα ως προτάσεις να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αν καθυστερήσουμε θα έχει δραματικές επιπτώσεις αυτό. Είμαι αισιόδοξο όμως και θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Θα λειτουργήσουν επικοδομητικά και θα τα πάμε καλά. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ήταν χθε, όχι, στι 19. 19 Δεκεμβρίου λοιπόν και θα έχουμε και συζήτηση σε σχέση με τις τροπολογίες. Θα γίνει στις 23 με 24 Ιανουαρίου αυτή η συζήτηση. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα συνέλθουμε στις 19 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε προ έγκριση και θα έχουμε την ψήφιση στην Ολομέλεια που δεν έχει ακόμα καθοριστεί ως ημερομηνία εξαρτάται από το πόσες τροπολογίες θα κατατεθούν από τους συναδέλφους σε σχέση με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση για τις επικοδομητικές προτάσεις, για τη θετική συζήτηση, για τις επικρίσεις αλλά και τις ε, θετικές παρατηρήσεις. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε το θέμα εδώ πάλι, το ETS, πάλι σύστημα εμπορίας ρήπων. Τι έχουμε εδώ, θέλουμε <clears throat> να μπορέσουμε το stop the clock, το θέμα δηλαδή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, υπευλήθη, η εδώ είναι ο Πέτερ Λίζε. Του δίνω αμέσως τον λόγο. Ως πρώτος θα παρέμβει ο Πέτερ Λίζε, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου μία εκπροημίου παρατήρηση ως προαπαιτούμενο, μια και τόσο ε, ζωηρά απευθυνθήκατε προς την κυβέρνηση του μεγαλύτερου κράτους μέλους προς την Γερμανία αληθεύει. Δεν έχουμε μια συντονισμένη θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας για το θέμα του backloading. Όταν όμως ε, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων συνήλθαν και με την Καγκελάριο, δεν ήταν τα πράγματα και τελείως διαφορετικά. Τώρα, για τις εναέριες μεταφορές εκπομπές ρήπων ε, θερμοκηπίου από τις εναέριες μεταφορές. Ε, μεγάλο μέρος ε, εδώ εμπλέκεται και, συμφων... και ομόφωνα αποφασίζεται προς αυτή την κατεύθυνση από το Συμβουλίο και είχαμε και μεγάλη πλειοψηφία. Ο πρόεδρος ήταν ο σκιώδης εισηγητής, εγώ ήμουνα ο εισηγητής ε, σε βάθος συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή Μεταφορών και τουλάχιστον από τη δική μου ε, κοινοβουλευτική ομάδα δεν είχαμε τροπολογίες, κανονική διαδικασία με πρώτη και δεύτερη ανάγνωση, δεν είχαμε τροπολογίες που να μην έχουν ε, συμφωνηθεί ή να έχουν συντονιστεί με τον εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών. Το λέω αυτό επειδή ο αξιότιμος εισηγητής της Επιτροπής Μεταφορών ανέφερε ότι ε, υπήρχαν ταλιμπάν λέει σε αυτή τη διεργασία. Ε, αυτά τα οποία όμως αποφασίσαμε, τα αποφασίσαμε από κοινού. Και δεν, είμαστε, δεν παρεκκλίναμε εμεί. Γιατί τα αποφασίσαμε. Επειδή οι εκπομπέ ρήπων στι ενέργειε μεταφορέ αυξήθηκαν και συνεχίζουν να αυξάνονται με δραματικού ρυθμού. Και επειδή και άλλοι φορεί μεταφορών στην συνεισφορά αυτή για την προστασία του περιβάλλοντο συνεισφέρουν, για παράδειγμα, τα ΙΟΤΑΧΗ και τα ε, φορτηγά οχήματα και σε πολλούς άλλους τομείς και οι σιδηρόδρομοι εντάσσονται στην ε, ε, πολιτική εκπομπών ρήπων. Δεν θα ήταν συνεκτικό τώρα οι εναέριες μεταφορές, τα αεροπλάνα να εξαιρούνται και σε σχέση με την ε, ιδιαίτερη επιβάρυνση μέσω των αερίων καυσαερίων τους που επιβαρύνουν το περιβάλλον να εξαιρούνται. Χάρη στο έργο που έγινε καταφέραμε με πολύ μετριοπαθή τρόπο, ε, τονίζω με μετριοπαθέστατες προτάσεις να εγκριθεί, να προχωρήσει η οδηγία. Στον τομέα της των εκπομπών ρήπων λέμε από το 2013 Κάνουμε λόγο για 21% μείωση σε σχέση με τις άλλες ε, βιομηχανίες. 5% ε, θα είναι στις ενέργειες μεταφορές ε, η μείωση. Η επιβάρυνση, πρέπει να το δούμε αυτό, σε σχέση με τις εκπομπές ρήπων, η επιβάρυνση θα είναι πολύ μετριοπαθής. Λέει στις διπυρωτικές πτήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα από το Λονδίνο προς τη Σανγκάη, 2 ευρώ. Στην ίδια την Ευρώπη η Ryanair ενδοευρωπαϊκά υπολόγισε ότι αν επιβάτη 25 σέντ θα καταβάλλονται, θα πρέπει να συνεισφέρονται ανά επιβάτη για διπυρωτικές ευρωπαϊκές πτήσεις. Αν δει κανείς τα μέτρα που κράτη-μέλη και τρίτες χώρες ε, ε, αποφάσαν, διανύμαμε ένα έγγραφο, ουσιαστικά θα έχουμε μια συζήτηση χωρίς έγγραφο, αλλά έχουμε και ένα προσωπικό έγγραφο δικό μου που έχει διανεμηθεί. Στη Γερμανία για διπυρωτική πτήση έχουμε 42 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανάλογα με την απόσταση και στην πρώτη θέση μέχρι 148 λίρες στερλίνες, πάνω από 200 ευρώ. Και στις ΗΠΑ υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση για διπυρωτικές πτήσεις 16 δολαρίων. Η Ινδία έχει 35 δολάρια ως ε, τέτοια επιβάρυνση. Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι αυτά τα οποία εγκρίναμε ήταν πραγματικά πολύ μετριοπαθή. Τώρα, υπάρχουν επικρίσεις έντονες από τρίτες χώρες Δυστυχώ, σχεδόν όλες οι τρίτες χώρε, οι ουσιοδέστερες τρίτες χώρε, με εξαίρεση την Αυστραλία και τον Καναδά που είναι μετριοπαθείς χώρες και που εργάζονται επικοδομητικά συνεργάζονται μαζί μας, η ΕΠΑ, η Κίνα όμως και η Ρωσία είναι μας δραστικά εναντίον αυτών των προτάσεων. Και τι γίνεται, έχουμε έξω εδαφική ε, ε, νομοθετική ισχύ σε τέτοιες ε, ρυθμίσεις και σε, στο έγγραφο αυτό βρίσκεται κάποιες πληροφορίες. Οι εθνικοί φόροι παρεκκλίνουν ανάλογα με την απόσταση. Αν από το Λονδίνο πάει κανείς στον Καναδά, πληρώνει κανείς ε, τη χαμηλότερη κλίμακα. Αν πετάει προς Μεξικό, υψηλότερη κλίμακα. Και βλέπουμε ενδιάμεσα έχουμε τη ΣΥΠΑ. Από την Γερμανία, Φραγκφούρτη προς Βαρσοβία, χαμηλότερη κλίμακα. Αν έχουμε Τόκιο, έχουμε υψηλότερη κλίμακα, διότι ενδιάμεσα βρίσκεται η Ρωσία. Το επιχείρημα δηλαδή ξαφνικά άρχισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει ρυθμίσεις και αποφάσεις που αφορούν τρίτες χώρες και μάλιστα άδικα, δεν μπορεί να ευσταθεί ένα τέτοιο επιχείρημα και το ΔΕΚ κιόλα είχε και μία προσφυγή αμερικανικών εταιριών την οποία πέριψε. Νομίζω ουσιαστικά υπάρχουν δύο επεξηγήσεις δύο ερμηνείες για αυτή την τεράστια αντίσταση, τεράστια πίεση από τρίτες χώρες. Πρώτον, σε τέτοιες τρίτες χώρες επικρατεί άποψη ότι εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν είμαστε σωστοί νομοθέτες, πραγματικοί αυθεντικοί νομοθέτες. Η άποψη επικρατεί ότι υπάρχει μια ιδέα λέει που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως στόχο και αν ασκηθεί πίεση παρεκκλίνουν οι ρυθμίσεις. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, ρυθμίσεις νομοθετικές που δεν, δεν ισχύουν και δεν ε, χρειάζεται κανείς να σέβεται. Αυτό είναι βέβαια προκατηλημένη άποψη των τρίτων χωρών και λυπούμαστε για το ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε δεδομένου αυτού. Το άλλο επιχείρημα όμως είναι πιο, ακόμα πιο ενδιαφέρον. Σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, το Υπουργείο Μεταφορών έχει τώρα την εντολή, αν δεν υπάρξει συμφωνία μαζί μας και, ε, παγκόσμια, αμερικανικές εταιρείε να απαγορεύεται να συμμετάσχουν στο σύστημα εμπορία τρύπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαν ε, οι υπεύθυνοι εδώ στι Βρυξέλλε και συζήτησαν μαζί μα έγιναν κιόλα μάλιστα υπήρξε και εκνευρισμό και υπήρξε και επιθετικότητα όταν εγώ ανέφερα το αμερικανικό νομοθέτημα Wexman Markey. Στο Κογκρέσο είχε σαφή πλειοψηφία, είχε την προσωπική υποστήριξη του Προέδρου Ομπάμα αυτό το νομοθέτημα. Απέτυχε δυστυχώ στην Γερουσία επειδή 60 ψήφοι που απαιτούντο δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν. Αυτό το νομοθετήμα προβλέπει εκπομπέ ρήπων για όλου του τομεί για τη βιομηχανία στη ΣΥΠΑ, παντού και για τι ε, μεταφορέ, ενέργειε μεταφορέ και για τι ε, κινέζικε και άλλε αυστραλιανέ και άλλε εταιρείε που εκκινούν από τη ΣΥΠΑ. Όταν ανέφερα αυτό το νομοθέτημα με παρεξήγησαν και εξοργίστηκαν αναφέρθηκε ότι το Wexman Mark είναι λέει θνησιγενές νομοθέτημα. Υπάρχει μια άλλη πλειοψηφία στο Κόγκρεσο και αυτή η νέα πλειοψηφία θα θέλει να μας καταδείξει ότι δεν είναι η ίδια όπως ήταν παλιότερα η περιβαλλοντική πολιτική από πλευρά στον ΗΠΑ. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα. Κάθε επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται ε, σε σχέση με το ETS θα μπορούσε και έναντι του Wexman Mark να αναφέρεται. Τα επιχειρήματα των Αμερικανών, ιδιαίτερα του Προέδρου Ομπάμα, είναι πολύ αποδυναμωμένα Ντροπή είναι η στάση του Ομπάμα. Πήρε το βραβείο Νομπέλ Ειρήνη, μεταξύ άλλων, και για τι προσπάθειέ του για την προστασία του κλίματο. Και τώρα υποβάλλει νομοθέτημα το οποίο ο ίδιο προσυπογράφει που το μόνο μέτρο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει το θέτει υποπίεση και το υπονομεύει. Έχουμε μια πολύ δυσχερή κατάσταση σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, διότι από όλε τι τρίτε χώρε ασκείται πολύ μεγάλη αντίσταση. Και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν είναι ότι θα θέλαμε να υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία και όχι, και όχι μια ευρωπαϊκή συμφωνία για παράδειγμα, που θα ρυθμίζει αυτά τα θέματα οικουμενικά. Εμείς απο, ε, καταστήσαμε σαφές ότι και εμείς θέλουμε μια οικουμενική, μια παγκόσμια συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι παγκόσμια από το 1997, από το το Κιώτο δεν έχει προχωρήσει καθόλου και δεν έχει αναλυθεί κάποια πρωτοβουλία. Τώρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι μια τέτοια διεθνή συμφωνία δεν θέλουμε να την παρεμποδίσουμε εμείς, αλλά σε περίπτωση που κάποιοι κολυσιεργούν είναι άλλοι και όχι οι Ευρωπαίοι. Και γι' αυτό είναι σημαντικό για την πρόοδο από πλευρά του ΑΙΚΑΟ, του πολιτικού οργανισμού αεροπορικών μεταφορών, μια ομάδα δημιουργήθηκε που θα μεριμνήσει ώστε το Σεπτέμβριο του χρόνου 2013, όταν θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση της ΑΙΚΑΟ, θα υπάρξει πρόταση προς λήψη απόφασης ε, ώστε να υπάρξει προώθηση μιας παγκοσμιοποιημένης τέτοια συμφωνίας. Κάθε τρία χρόνια συνέρχονται στην Ολομέλειά του και τώρα θα είναι πραγματικά η ευκαιρία να υποβληθεί πρόταση για την επίλυση του προβλήματο. Διαφορετικά θα χάσουμε πάλι τρία χρόνια, δεν θα γίνει τίποτα για τρία χρόνια. Υπό αυτό το σκηνικό πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει το χρονόμετρο και να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τη δική μας οδηγία που θα ε, ετίθετο ε, εκτός δεν θα εφαρμοζόταν για ένα χρόνο. Θα πρέπει να δούμε αν αυτό μπορεί να γίνει και είναι σωστό. Πρώτες σκέψεις είναι ότι με μια πρώτη αξιολόγηση μπορούμε να πούμε ναι. Έκανε ένα FES, μια ευφυή κίνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποδείξουμε ότι δεν κολλησιεργούμε έναν μια παγκόσμια συμφωνία. Αν λειτουργήσουν τα πράγματα, τέλεια. Θα έχουμε αυτή την κατάσταση που επιθυμούμε. Αν δεν λειτουργήσουν, θα είναι σαφέ ότι δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι δεν επετεύχθη μια παγκόσμια συμφωνία. Και έτσι, σε σχέση με τι ενέργειε μεταφορέ, μπορεί η πίεση να πάψει να εφαρμόζει να ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν θα φταίει εκείνη για τους συναδέλφους που ε, θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε σχέση με αυτή τη συζήτηση επί των προτάσεων που κατατίθενται. Υπάρχουν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει διαφορά διπυρωτικών πτήσεων και ενδοευρωπαϊκών πτήσεων. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμφωνία να ισχύει μόνο, να, να πάψει να ισχύει μόνο, να εξαιρεθεί μόνο για διπυρωτικές πτήσεις διότι ε, σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες εμείς δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο μονομερός αλλά να γίνουν και τα δύο και να δούμε δεδομένη της νέας κατάστασης τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Έχει προτερήματα και μειονεκτήματα η κατάσταση αυτή. Θα έλεγα να μην αναμείνουμε τα πράγματα. Κάθε τροποποίηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεπάγεται προβλήματα και περαιτέρω συζητήσεις. Πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι του χρόνου πριν από το καλοκαίρι μέχρι το Μάιο για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Να δούμε την πρόταση. Τι θα γίνει με τις ε, παρόχους πτήσεις, ε, ε, πτήσεις ανταποκρίσεις που οδηγούν επιβάτες από ένα μικρότερο αεροδρόμιο σε ένα μεγαλύτερο αεροδρόμιο και από εκεί ξεκινούν οι διπυρωτικές πτήσεις νωρίτερα και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εταιριών εναέριων μεταφορών για να προστατευτούν από αθέμητο ανταγωνισμό από έξω ευρωπαϊκές εταιρείες υπάρχει πρόταση αυτές οι πτήσεις ανταποκρίσεων να εξαιρεθούν και αυτές για ένα χρόνο. Είναι πάρα πολύ ε, ακαθόδες το θέμα και δύσκολο. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τελευταίο σημείο που πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εξειδικευθεί είναι να δούμε τι αναμένουμε ακριβώς, τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο. Μπορώ να προβλέψω και να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο 2013 δεν θα έχουμε μια λύση που θα μας ικανοποιεί όλους και θα ισχύσει άμεσα. Όχι, καθόλου. Θα έχουμε μάλλον μια λύση, αν είμαστε τυχεροί και αν έχουμε κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις μας, μια λύση που θα αρχίσει να εφαρμόζεται και να ισχύει μετά από μερικά χρόνια δεν θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2013 μια παγκοσμιοποιημένη τέτοια συμφωνία όπου ικανοποιητικά θα έχουν ρυθμιστεί οι εκπομπές ρήπων ε, από τις εναέριες μεταφορές σε ένα έγγραφο ερωτήσεων απαντήσεων, questions and answers, που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α, παρουσιάζει το τι αναμένει εκείνη, αλλά δεν είναι νομοθετική πρόταση. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια συμφωνία που θα βασίζεται στι αγορέ, δηλαδή ένα σύστημα εκπομπών ε, ε, ρήπων ή κάτι παρόμοιο, ώστε να συμμετάσχουν όλοι. Και αν αυτό δεν ισχύσει από την 1η Πρώτου 2014, τότε για τη μεταβατική περίοδο χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα έχει ένα σύστημα τροποποιημένο που θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί είναι σαφές, δεν μπορούμε επειδή υπόσχεται η ICAO ότι το 2020 θα κάνει ίσως κάτι λέει, μέχρι τότε να μην κάνουμε εμείς τίποτα και να καταργήσουμε τις ρυθμίσεις μας. Θα πρέπει για τη μεταβατική περίοδο να γίνουν τα αναγκαία βήματα και διαβήματα που θα μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την αναγκαία πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πέτρα Λίζε και προαναφέρθηκε αυτό. Εγώ ήμουν σκιώδης εισηγητής για αυτό το θέμα, για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Προτού τώρα θεματολογικά ε, αρχίσουμε τη συζήτηση, θέλω ένα υπουργό να χαιρετήσω. Από το ε, Βάλις ε, Καλώς ήρθατε την Ουαλία. Καλώς ήρθατε λοιπόν Ουαλέ Υπουργέ Μεταφορών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Όσον αφορά την πρόταση αυτή, Ευραίω και διεξοδικά συζητήσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε δύο αναγνώσεις για αυτή την πρόταση και ήταν μια συμβιβαστική πρόταση αυτή. Ρητά ένας συμβιβασμός μεταξύ των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και των μελών της Επιτροπής Μεταφορών. Ο πιστοδρομήσαμε σημαντικά και υπήρχαν πολύ μεγάλες επιφυλάξεις αν διεθνώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όλα αυτά. Τώρα, η οργάνωση για τις ε, διεθνείς αερομεταφορές, ε, η ΑΟΚΑΟ, συζητά αυτή η οργάνωση από το 13-14 χρόνια σχεδόν κιόλα, Πώς σφαιρικά, συνολικά μπορεί να θεσπιστεί, να εισαχθεί ένα σύστημα για την προστασία του περιβάλλοντος και διεθνώς να ρυθμίζεται ένα τέτοιο σύστημα. Βλέπουμε ακριβώ στην Ευρώπη και ο Πέτερ Λίζε το προανέφερε ότι η αγορά έχει κατακαιρματιστεί συνολικά. Έχουμε διαφορετικούς φόρους, διαφορετικά τέλη. Στην Ολλανδία υπήρχε ένα τέλος. Υπήρξαν όμως κάποιοι ευφυεί επιχειρηματίες που κοινούσαν κινούσαν επιβάτες με λεωφορεία, με πούλμαν. Ήταν πλήρη αυτά τα πούλμαν τότε. Τώρα εισήχθη ένα τέτοιο τέλος στη Γερμανία και κινείται αντίστροφα αυτή η ροή τώρα. Δηλαδή όλα αυτά που θέλαμε να εντάσσονται σε μια ενιαία εσωτερική αγορά δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Και η πρόταση που έχουμε εμείς που προχώρησε, δηλαδή οι εναέριες μεταφορές να ενταχθούν στο εμπόριο εκπομπών ρήπων και οι εξωτερικές πτήσεις επίσης ήταν η σωστή προσέγγιση όμως τα κράτη-μέλη πρέπει να μεριμνήσουν να λειτουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Είτε εκπομπές ρήπων είτε τέλος που θα επιβάλλεται. Και τα δύο δεν μπορούν να λειτουργήσουν αμφότερα. Είμαι υπέρμαχος νομοθετικής ρύθμισης εγώ. Θερμός υπέρμαχος. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταματήσει το χρονόμετρο, δηλαδή να πάψουν να ισχύουν κάποιες ρυθμίσεις για ένα χρονικό διάστημα έχουν συζητηθεί και με τον, Υπουργό, ε, τον Κινέζο Υπουργό. Τα μηνύματα που είχαμε από οι Άπωνες συναδέλφους και από άλλους ήταν πρέπει να πω θετικά τα περισσότερα. Πρέπει να είναι όμως σαφές ότι επί της ουσίας θα δημιουργούν ένα συγκρίσιμο πλαίσιο σε ένα επίπεδο συγκρισιμό, συγκρισιμότητας διεθνώς αν κάνουμε αυτό το βήμα και προχωρήσουμε και να μην υπάρχει κατακαιρματισμός. Υπάρχουν συμπάθειες λοιπόν με αρκετή κατανόηση αντιμετωπίζουν αυτή την προσέγγιση και από πλευράς Επιτροπής ε, είχαμε και την ε, αντίστοιχη τέτοια αντιμετώπιση. Αν όλα αυτά είναι δυνατόν να γίνουν διεθνώς να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία που να έχει αυτή την ουσία δεν μπορεί να είναι πρόσχημα ή να είναι μια δικαιολογία. Αν όμως δεν πετύχει αυτό, αν όλα αυτά ευδοκιμήσουν θα μπορέσουν να ανοίξουν οι δυνατότητες για να λειτουργήσουν τα πράγματα και αλλού. Και στην Κίνα γίνονται πράγματα. Και σε επτά περιφέρειες ε, της Κίνας άρχισε ένα τέτοιο σύστημα εκπομπών ρήπων. Προβλέπεται η ένταξη όλης της Κίνας, του συνόλου της Κίνας σε αυτό το πλαίσιο. Από πλευράς είπα η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Μπορεί κανείς να δει τα πράγματα ότι δεν θέλουν να περάσουν σε μια διαπραγμάτευση χωρίς να έχουν επιρροή, χωρίς να έχουν μοχλική ε, επιρροή. Γι' αυτό είμαι προσεκτικά αισιόδοξο όσον αφορά την κατάσταση στην ΑΙΚΑΟ θα έπρεπε πιστεύω να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία που μόλις διαγράφησε και ο εισηγητής. Δηλαδή να υπάρξει μια εξαίρεση των διεθνών πτήσεων. Όχι των διευρωπαϊκών πτήσεων, αλλά των διεθνών διπυρωτικών ε, πτήσεων. Εμείς στις διευρωπαϊκές πτήσεις έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία. Εγώ στη βορειοδυτική μας περιοχή στη Γερμανία έχουμε και νησιά όταν θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια διαδρομή πληρώνουμε κάτι παραπάνω για τα ανατολικά νησιά της Φρισλανδίας για παράδειγμα σε σχέση με την διαδρομή ε, προς Washington δηλαδή τριπλό, τριπλή επιβάρυνση όσον αφορά το τέλος αυτό η αναλογικότητα του όλου θέματος. Πώς δηλαδή αντιμετωπίζεται θα έλπιζα να ίσχυε και στη συζήτηση για το τέλος για το διοξίδιο του άνθρακα στις χώρες μας διότι υπάρχουν σημαντικές παρεκκλήσεις και αυτές οι κινήσεις μεταξύ των κρατών μελών δηλαδή κάποιοι να μετακινούνται με πούλμαν και να πηγαίνουν στο πιο κοντινό αεροδρόμιο αυτό είναι ένα μέσο παρέκκλησης. Πρέπει να δούμε ότι η συνολική εμπορία ρήπων πρέπει να λειτουργήσει. Με την ένταξη στο πλαίσιο τρύπων και των εναέριων μεταφορών. Αυτή την ευκαιρία πρέπει να εκμεταλλευτούμε τώρα και έτσι να δράσουμε και να πούμε κάθετα και με σαφήνεια ότι στις 31 Δωδεκάτου αν δεν γίνει τίποτα μέχρι τότε εμείς θα συνεχίσουμε με το νομοθετικό μας έργο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να εξακολουθήσει να υφίσταται η πίεση, νομοθετική πίεση κίνησης, να κινητοποιηθούν κάποιοι προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπω συγκατανεύετε εσείς συνάδελφε Φώστερ, να μην δηλαδή απεμπολίσουμε εδώ τα δικαιώματά μας, να ασκήσουμε την επιρροή μας, να έχουμε μόχλευση ώστε να ασκήσουμε την επιρροή μας. Υπό όρους και προϋποθέσεις, όχι χωρίς και προϋποθέσεις Davis όμως. Επόμενος σκιώδης εισηγητής, Chris Davis. Παρακαλώ. Thank you. Thank you, Chairman. And, uh, and thank you Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ βέβαια και τον uh, Πίτερ ε, Λίζε ε, γιατί ξέρουμε ότι ασχολείται πολλά χρόνια με τα θέματα αυτά και της αεροπορίας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί θέλουμε να συμπεριληφθεί εδώ και η αεροπορία. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί μια και έχουμε πρόσφατη τη συζήτηση για την Τόχα, νομίζω ότι εδώ εντάσσεται πάρα πολύ καλά το ζήτημα και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να παίξει ηγετικό ρόλο, προσπάθησε να είναι καινοτόμα και, και με αυτό τι, τι κατάφερε πολύ λίγα ένα από τα θέματα της αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή είναι ότι κάθε χώρα στον πλανήτη έχει ε, ε κοινέ ε, ευθύνες αλλά λίγο διαφοροποιημένες. Το θέμα είναι ε, να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνονται τη στιγμή που πρέπει και αυτό πρέπει να κάνουμε από την αρχή έγινε σαφές και από την Κομισιόν και από άλλους ότι ε, ε, το ε, ζήτημα ήταν να έχουμε διεθνείς συμφωνίες όσον αφορά τις εκπομπές ε, που παράγονται από, την, ε, από τις αεροπορικές μεταφορές. Ε, ο κόσμος το αναγνωρίζει ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ προσπαθούμε να πιέσουμε όλους έτσι ώστε να γίνει και κάτι και στην πράξη και όχι μόνο να ανταλλάσσουμε λόγια. η Κομισιόν ε, χρησιμοποίησε την εφαρμογή του ETS για να πιέσει ε, κάποια συζήτηση και κάποια έτσι πρόοδο. Η Κομισιόν ήρθε και σε εμά και είπε ότι πιστεύει ότι έχει ήδη γίνει σημαντική πρόοδος ε, και βεβαίως υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, αλλά πάντα γίνεται αυτό όταν δρά με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι γενικώ υπάρχει μια καλή πρόοδος ε, και ότι ε, με τον τρόπο αυτό και μάλλον και οπισθοδρομεί λίγο έτσι ώστε να δώσει περισσότερο χώρο για διαπραγματεύσεις. Και μας λέει και το το χρονοδιάγραμμα ε, είναι τέτοιο που δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συμφωνία πριν από το ε, ETS ε, και ζητάει λίγο χρόνο και μας λέει στηρίξτε με στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως ε, επικρίθηκε τα μάλα από τους πρασίνους και από κάποιους από τη δικιά μου ομάδα ότι δεν τα έκανε καλά, ότι δεν ήταν αρκετά, ε, ε, δεν υπήρξε πρόοδος, ότι δεν ήταν αρκετά φιλόδοξα τα προγράμματα. Κάποιοι άλλοι από άλλες πολιτικές σκοπιές δεν συμφωνούσαν και επέκριναν την ιδέα, τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, ήθελε η Κομισιόν ε, να πιέσει ας πούμε τη συζήτηση. Δηλαδή στην ουσία βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι ε, δεν θέλει να προχωρήσει στη δέσμευσή τη ε, η Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι κανεί το πιστεύει εδώ. Γι' αυτό λοιπόν α προσπαθήσουμε να αφήσουμε τα πράγματα απλά. Α προσπαθήσουμε να μην προσθέτουμε πράγματα. Να στηρίξουμε την Κομισιόν στο διαπραγματευτικό τη ε, ρόλο και νομίζω ότι όσο πιο ενωμένοι είμαστε και όσο πιο απλοί είμαστε, τόσο πιο ε, στεναρό είναι και το μήνυμα που στέλνουμε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να είμαστε αυστηροί, ότι το ETS θα εφαρμοστεί ε, στα ε, ευρωπαϊκά αεροδρόμια τουλάχιστον εάν δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία και αυτό πρέπει να είναι σαφές και κατανοητό από όλους. Και επίσης ότι βεβαίως θα πρέπει στην ΑΙΚΑΟ να γίνει στη Γενική Συνέλευση να γίνει πρόοδος. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστ. Και τώρα Φώστερ, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Έχετε δίκιο πρέπει να μετριάσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλη την υποστήριξή μας. Εξετάζουμε τον νέο ευρωπαϊκό ουρανό, τις πρόοδους της τεχνολογίας. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε υποστηρίξει τον καθαρό ουρανό, την καθαρή τεχνολογία. Κατά... Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε. Το δύσκολο εδώ και αυτό δεν είναι λάθο ούτε των μελών αυτή τη Επιτροπή, ούτε των μελών τη Επιτροπή ε, Μεταφορών. Είναι ότι αυτή η πρόταση είχε κάποιο ελάττωμα. Σταθερό καθεστώς για το, ε, την ανταλλαγή εκπομπών, γιατί δεν μπορεί εκπομπών, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν το πρότεινε η Κομισιόν πριν από μερικά χρόνια, δεν είχε προβλέψει ότι θα υπάρχουν πάντα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα με τρίτες χώρες, νομικά ζητήματα σε θέματα με την επιβολή φόρων σε μεταφορείς τρίτων χωρών. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν μας άκουσε για αυτό το θέμα. Ακούσαμε και άλλε πολλέ διαφορετικέ απόψει από νομικού συμβούλου που είπαν ότι δεν πρέπει να προχωρήσετε προ αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, εδώ είμαστε τώρα και τώρα τα πράγματα έχουν γίνει άνω κάτω. 170 χώρε όταν το προτείναμε αυτό ε, είπαν στην Κομισιόν ότι έχουμε προβλήματα. Τώρα έχουμε μεγάλε σημαντικέ χώρε, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, που έχουν νομοθεσίε στι δικέ του χώρε όπου οι εταιρείε του, βάσει τι οποίε οι εταιρείε του δεν μπορούν να συμμορφωθούν με αυτό το σύστημα εμπορία ε, ε, ε, ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τώρα διαφορετικέ θέσει, διαφορετικέ απόψει. Άλλα κράτη-μέλη θέλουν να προχωρήσει, άνθρωποι σαν εμένα πιστεύουμε ότι δεν είναι ίσω στην κατεύθυνση. Και τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία stop the clock. Τι σημαίνει stop the clock, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται οι μεταφορέ των τρίτων χωρών, αλλά από την Κομισιόν μου είπαν πριν μερικού μήνε θα πρέπει να αναβληθεί για όλου αν είναι να αναβληθεί οι μεταφορεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δικές μας επιχειρήσεις, τους επιβάλλουμε ένα φόρο, ενώ δεν επιβάλλουμε τον φόρο αυτό σε ε, εταιρείε τρίτων χωρών, τις οποίες ουσιαστικά αφορούσε αυτός ο κανονισμός. Έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας εδώ πέρα, διότι τι κάνει η Κομισιόν, έρχεται και μας προτείνει έναν κανονισμό, τα κράτη-μέλη πολύ σωστά συμμορφώνονται, τον εντάσσουν, τον μεταφέρουν στην νομοθεσία τους και μετά οι μισή από εκείνους που θα εμπλέκονταν σε αυτό δεν το υλοποιούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να λέμε για το μετριασμό των εκπομπών και όλα αυτά. Τώρα η ΚΑΟ είναι η απάντηση. Η ΚΑΟ θα συνεχίσει να λέει διάφορα, αλλά δεν, έχει, δεν μπορεί να επιβάλλει κάποια νομοθεσία. Ως οργανισμός είναι ένα σώμα όπου ελπίζουμε ότι διάφοροι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποφασίσουν να υλοποιήσουν κάτι. Κατά την άποψή μου, εδώ μιλάμε να σταματήσουμε το ρολόι, να σταματήσουμε το ρολόι σε ποιο πράγμα. Τι θα συμβεί σε 12 μήνες όταν οι τρίτε χώρε ε, που ε, ψήφισαν νόμου μη συμμορφώσει των εταιρείων τους με αυτό το κανονισμό συνεχίσουν να εφαρμόζουν την ίδια μη συμμόρφωση. Τι θα κάνουμε τότε για να είμαστε ρεαλιστές και να είμαστε δίκαιοι προ του ε, Ευρωπαίου αερομεταφορεί, θα πρέπει να αναστείλουμε το όλο ζήτημα και μετά να δούμε τι μπορούμε να επινοήσουμε αλλά το να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό που έχει ουσιαστικά καταρρεύσει κανείς δεν άκουσε αρχικά τις απόψεις που έλεγαν ότι αυτή δεν ήταν η απάντηση για το μετριασμό των ρήπων. Ήταν υπερβολικά περιοριστική η πρόταση αυτή, ήταν υπερβολικά γραφειοκρατική και έτσι φτάσαμε εδώ που είμαστε με το να μην ακούει η Κομισιόν τι διάφορε συμβουλέ και τώρα έρχονται και μα λένε λύστε το. Ε, δεν το ξεκινήσαμε εμεί αυτό. Δεν ήταν η Επιτροπή Περιβάλλοντο, ούτε η Επιτροπή Μεταφορών που το ξεκίνησε ή το πρότεινε αυτό. Η Κομισιόν το πρότεινε και η Κομισιόν δυστυχώ τώρα μα ζητάει να του σώσουμε, να του διασώσουμε και η δική μου πρόταση δυστυχώ θα ήταν, ήταν, αν θέλετε να το αναστείλετε, αναστείλτε το. Και μετά ελάτε σε εμά κάποια στιγμή στο μέλλον και πείτε μα η ΚΑΟ δεν βρίσκει άκρη, α ξεκινήσουμε από την αρχή. Το να κάνουμε stop the clock, όπω λέτε, να σταματήσουμε το ρολόι, δεν νομίζω ότι αυτή είναι καλή απάντηση. Εγώ προσπαθώ να υποστηρίξω τη δική μου βιομηχανία, το δικό μου τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλω να ανταγωνίζονται παγκοσμίω με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη. Γιατί να πληρώνουν φόρου που δεν θα πληρώνουν οι τρίτε χώρε, επειδή εσεί ψηφίσατε, προτείνατε μάλλον, ελλειπή νομοθεσία ευθύ εξ αρχή. Αυτά έχω να πω εγώ και θα με ενδιαφέρει να δω τι θα μα αναφέρει σήμερα η Κομισιόν. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό και στην Επιτροπή Μεταφορών πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λίντα Μακέβαν. Τι να σας πω να πω στην Τζάκη Φώστερ ότι έκανε μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτοί που ενέκριναν αυτές τις προτάσεις, αυτή την ομοθεσία, πέρασε από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού, δηλαδή από βουλευτές και ε, υπουργούς. Εν πάση περιπτώσει ε, και ε, στην τελευταία Βουλή οι εκπρόσωποι του κόμματός σας είχαν στηρίξει αυτή την νομοθεσία. Ε, και επομένως να μην λέμε και πολλά. Δεν είναι ανόητη αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως μερικοί θέλουν να την παρουσιάζουν και πρέπει κάπως να στηρίξουμε και την Κομισιόν. Να πω στους εκπροσώπους ε, της Κομισιόν ότι με αγχώνει λίγο αυτή η πρόταση, πέρα από όσα είπε η Τζάκι Φώστερ είναι ότι όσοι αντιτίθεντο σε οποιαδήποτε δράση κατά της ε, ε, συμπερίληψης της αεροπορίας ε, τώρα βρίσκουν μια εξαιρετική ευκαιρία να σταματήσουν την ε, διαδικασία. Ξέρετε ότι αυτό το τέλος είναι πολύ μικρότερο σε σχέση ε, με τα ε, τέλη που εφαρμόζουν κάποιες κυβερνήσεις και ο, ξέρετε, 8 λίρες τερλίνες αναπόδι είναι για τις υπερατλαντικές πτήσεις η χρέωση. Εάν η ΚΑΟ δεν προτείνει είναι γιατί και εμείς δεν είχαμε από την Κομισιόν καμία πρόταση. Δεν ε, είδαμε ούτε στο, ε, στον IMO οποιαδήποτε πρόοδο όσον αφορά τις θαλάσσιες εκπομπές γιατί δεν υπήρχε πίεση από τον IMO. Δεν, δεν είχε πίεση μάλλον ο IMO. Είχαμε πριν από λίγους μήνες τη συζήτηση για το ETS, μόλις είχαμε μια άλλη συζήτηση, είχαμε ε, και ε, ε, κάποια που έκαναν έτσι πολύ, άσκησαν πολύ μεγάλη πίεση, έκαναν μεγάλο λόμπι, λόμπι και ξανανοίξαμε και την οδηγία για τα καλλιντικά και νομίζουν μερικοί ότι διαρκώς μπορούν να, ακολουθούν την ίδια τακτική. δεν μπορούμε όμως, γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε σοβαροί όσον αφορά την κλιματική αλλαγή θα μπορούσα να συμφωνήσω με τον Chris Davis, ε, δηλαδή ε, να πούμε ότι ε, συμφωνούμε με μια γρήγορη διαδικασία, αλλά η ανάκληση της νομοθεσίας να μην είναι διαρκής Δηλαδή, εάν δεν προχωρήσει το πράγμα, τότε αυτομάτως να εφαρμοστεί ε, η νομοθεσία. Και αυτή είναι η ερώτηση προς την Κομισιόν. Πότε θα ξέρουμε, ποιος θα, κάνει, ποιος θα αποφασίσει αν η πρόταση της ΙΚΑΟ είναι σωστή ή όχι, είναι καλή ή όχι. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο, πόσο αυτόματη θα είναι η διαδικασία και πώς ε, προχωράει η συζήτηση στο Συμβούλιο, κυρίως ε, από τις χώρες που δεν θέλουν καμία συμφωνία στην ΙΚΑΟ. από ό,τι βλέπουμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν προβλέπουμε και μεγάλη στήριξη από τις ΗΠΑ. Ε, θα θέλαμε κάποια σχόλια όσον αφορά το τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ξανανοίξαμε λοιπόν την, ε, τον νόμο πριν από λίγο και οι περισσότεροι από εμά τότε είχαν την αίσθηση ότι δεν έπρεπε να ξανανοίξει το ζήτημα αυτό, αλλά ξανάνοιξε και το συζητάμε. Και ελπίζω να μην ε, καταστρέψουμε οποιαδήποτε ελπίδα είχαμε για ρύθμιση των εκπομπών στην αεροπορία τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Φρανσουάς Γκροστέτ. Ε, συγγνώμη, περιμένω να τελειώσει και η διερμηνία να, να ακούσω το σύνολο. Ωραία, όσον αφορά αυτό το ζήτημα το οποίο είναι ε, σημαντικό αλλά το συζητάμε διαρκώς, ε, είναι ο ρόλος της αεροπορίας στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Μπορώ να συμφωνήσω επί της αρχής, αλλά ε, όσον αφορά την υλοποίηση, αυτή προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Γιατί αν δημιουργήσουμε νομοθεσία μόνο για την Ευρώπη, τότε όντως δημιουργούμε προσκόμματα και δυσκολίες στις, ε, στους αερομεταφορείς μας. Θα θέλαμε μια διεθνή συμφωνία. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς Ευρωπαίοι. Χρειαζόμαστε αυτή τη διεθνή συμφωνία, γιατί διαφορετικά τότε τότε οι αεροπορικές μας εταιρείες θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, σε άσχημη ανταγωνιστική θέση και θα προλιάνουμε το έδαφος ε, για ε, την, ε, για την αεροπορική μας αγορά. Ξέρετε ότι έχουν ήδη παγώσει ας πούμε οι παραγγελίες Airbus και πηγαίνουν προς την Κίνα. Βεβαίως εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε κατά της κλιματικής αλλαγής αλλά χωρίς να αυτοπυροβολούμαστε γιατί διαφορετικά τίποτα δεν θα γίνει σωστά. Χαίρομαι που η ε, Επίτροπος που είναι υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή έχει αναβάλει την εφαρμογή αυτού του ε, τέλους για την ώρα γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτή τη διεθνή συμφωνία γιατί διαφορετικά δημιουργούμε προσκόμματα στις ίδιες μας τις αεροπορικές εταιρείες. Εγώ θέλω να προχωρήσουμε με εξαιρετικά μεγάλη σύνεση και προσοχή. Εγώ θέλω ε, να πω ότι είμαι και πολύ προσεκτική αλλά και ιδιαίτερος διστακτική όσον αφορά αυτό το δασμό. που έχει μετατεθεί χρονικά και θα πρέπει να εργαστούμε σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Για μπράτη, παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που έχουν ήδη πει οι συναδελφοί μου. Αλλά ας το συμφωνήσουμε καθαρά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε για οποιαδήποτε μέτρα καταπολέμησης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι το όλο ζήτημα του ισότιμου ανταγωνισμού. ο τομέα, ε, όπου έχουμε αυτόματο ισότιμο ανταγωνισμό είναι η αεροπλοεία, διότι εκεί φορολογούμε όλες τις εταιρείες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είμαι λοιπόν απόλυτα πεπισμένος ότι το ζήτημα εδώ δεν είναι τα πρακτικά προβλήματα. Εδώ μιλάμε για ζήτημα αρχής. Οι περισσότερες χώρες και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να φορολογηθεί η αεροπορία. Το είδαμε με την κεροζίνη, με όλα τα ΦΠΑ που σχετίζονται με την αεροπορία. Δεν υπάρχουν. Ας είμαστε λοιπόν ειλικρινεί σε αυτή τη συζήτηση και όχι να παρουσιάζουμε περίεργα επιχειρήματα. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Εάν το ζήτημα εδώ ήταν ο ανταγωνισμός, θα μπορούσε να είναι. Πώς είναι δυνατόν να είναι ζήτημα ανταγωνισμού όταν ένα φλιτζανί καφέ στο αεροδρόμιο του Χίθρου είναι πιο ακριβό από το φόρο που πληρώνω για να πάω στη Σαγκάη. Δηλαδή μου κοστίζει 2 ευρώ. Ποιο σε αυτόν τον κόσμο θα αλλάξει αεροπορική εταιρεία για διαφορά 2 ευρώ. Δεν νομίζω ότι κάποιο θα το κάνει. Στη μια αεροπορική εταιρεία, σε μια αεροπορική εταιρεία όπου παίρνεις ε, τα ποτά σου τσάμπα θα συνεχίσει. δεν θα έχει σχέση με τη φορολόγηση αυτό. Δηλαδή η ερώτησή μου προ την Κομισιόν είναι το ζήτημα εδώ είναι ανταγωνισμό ή απλά ότι δεν θέλουμε να αγγίξουμε την αεροπορία καθόλου. Εκεί στο πολιτήριο όπου 2 ευρώ δίνουν καφέ στο Χήθρο θα ήθελα να μου την δείξετε. Πού είναι αυτό το καφενείο για 2 ευρώ καφέ στο Χήθρο. Πρωτού όμως ο συνάδελφος Γιαμπράντη μου δείξει αυτό το πολιτήριο θα δώσω τον λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Πράγματι, τα σχόλια σας τα... μας βοήθησαν ιδιαίτερα να καταλάβουμε τόσο την υποστήριξη όσο και τις ανοιχτές ερωτήσεις, τις εκκρεμούσες ερωτήσεις που απομένουν όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν ανέκαθεν ήταν και παραμένει υποστηρικτή των καθολικών λύσεων, των οικουμενικών λύσεων. Από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία των 97, συμμετείχαμε και συμβάλαμε ενεργά σε αυτές τις συζητήσεις. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία ΚΑΟ, δεν έχει παρέχει έγκαιρα αποτελέσματα για δράση που να έχει νόημα. Γι' αυτό το λόγο έκανε την πρόταση της Επιτροπή να συμπεριληφθεί η αεροπορία στο ETS από το 2012. Εμείς κατά κανένα τρόπο δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, ότι τα μέτρα μας δεν είναι νόμιμα. Η νομιμότητα έχει αποδειχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έγινε ευρεία δημόσια διαβούλευση που οδήγησε στην υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που περιλαμβάνει την αεροπορία στο ETS. Και αυτό δεν είναι νομοθεσία της Κομισιόν, είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους τους ενδιαφερομένους που εμπλέκονται στις τρέχουσες αποφάσεις και συζητήσεις για λήψη αποφάσεων. Γιατί λοιπόν αυτό παραμένει το κεντρικό σχέδιο για την παροχή οικουμενικής λύσης. Είναι σαφές από, από τότε που συμπεριλήφθη το EU ETS, το ETS οι πρόοδοι επιταχύνθηκαν. Είναι άνευ προηγουμένου το ότι καθιέρωσαν ομάδε εμπειρογνωμών που αφιέρωσαν πόρου και χρόνου συνεδριάσεων να συζητήσουν και να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα των ε, μέτρων που βασίζονται στην αγορά. Και αυτά τα μέτρα δεν είναι μόνο το ETS. Είναι διάφορα καθεστώτα αντιστάθμισης που εξετάζονται κάποια σε σχέση με έσοδα, κάποια άλλα χωρίς. Το Συμβούλιο της 9ης Νοεμβρίου συμφώνησε ότι αυτά τα μέτρα τεχνικά είναι εφικτά, είναι υλοποιήσιμα, αλλά χρειάζεται να έχουμε μια συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο ώστε να διευκολυνθεί η οθέτηση αυτών των μέτρων. Για να διευκολυνθεί λοιπόν αυτή η πολιτική διαδικασία, μια ομάδα υψηλού επίπεδου συγκροτήθηκε από τον πρόεδρο Κομπέ υπό την προεδρία του και συναντήθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά ώστε να, παρέχει, να παρέχει πολιτική καθοδήγηση η οποία έλειπε από τις τεχνικού τύπου συζητήσεις για τα διάφορα καθεστώτα που βασίζονται στην αγορά. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που ανέφεραν ότι είναι απίθανο ένα οικουμενικό ενιαίο μέτρο να μπορέσει να υιοθετηθεί και να τεθεί σε λειτουργία από τότε που μετά τη συνάντηση το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του επόμενου έτου τη ΣΥΚΑΟ, τη συνέλευση τη ΣΥΚΑΟ. Αλλά αυτό που είναι δυνατό είναι η καθιέρωση ενό πλαισίου μέτρων που θα επιτρέψει την ύπαρξη εθνικών και περιφερειακών μέτρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή και να ανοίξει ο δρόμος για την ενδεχόμενη υιοθέτηση πραγματικά ενό οικουμενικού, ενό καθολικού ενιαίου μέτρου. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεδομένη τη προόδου που σημειώθηκε στη συνάντηση του Συμβουλίου τη 9η Νοεμβρίου, η Επιτροπή πρότεινε στι 12 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά να εφαρμόσει εξαίρεση στην εφαρμογή του ETS για την αεροπορία όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές εντός προς την Ευρώπη και που βγαίνουν εκτός Ευρώπης. Αυτή η εξαίρεση ισχύει, ισχύει για όλες τις ε, αεροπορικές εταιρείες ανεξαρτήτως εθνικότητας. Όταν πετάει η Lufthansa από τη Φραγκφούρτη στη Washington, εξαιρείται από το μέτρο. Όταν πετάει η British Airways από το Heathrow στη Νέα Υόρκη, εξαιρείται. Αν όμως η Air China πετάει εντός της Ευρώπης, τότε καλύπτεται, ε, ισχύει για αυτήν η νομοθεσία. Οι τρίτες λοιπόν, οι τρίτων χωρών μεταφορής οι μεταφορές τρίτων χωρών πρέπει να συμμορφώνονται για εγχώριες πτήσεις. Το stopping the clock ουσιαστικά αφαρμόζει αρχές μη διάκριση στο πλαίσιο του ETS και διαβεβαιώνει, διασφαλίζει ε, συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες. Αυτή την πρόταση δεν την επινοήσαμε εμείς ε, εκ του μηδενός. Τη μελετήσαμε προσεκτικά, την αξιολογήσαμε από απόψη σκοπιμότητας, υλοποιησιμότητας, πρακτικής δυνατότητας εφαρμογής. Μην, κάνετε, μην απατάστε. Οι αερομεταφορείς μας, οι αερομεταφορείς τρίτων χωρών, καθώς και τα κράτη-μέλη που διαχειρίζονται την εφαρμογή του ETS για την αεροπορία χρειάζονται σαφήνεια. Πρέπει να μπορούν να δράσουν εκ των προτέρων, προβλέποντας μια συμφωνία. Όσο πιο σαφή είναι η απόφαση, τόσο πιο σαφέ θα είναι το ETS και η διαστάσει του για τον υπόλοιπο κόσμο. Αληθεύει ότι οι συνάδελφοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπούν εμά στι ε, διαβουλεύσει ομάδων υψηλού επίπεδου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν αυτέ τι συζητήσει από ευρωπαϊκή προοπτική ώστε να υπάρχει κάποια μόχλευση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ε, τα χρονοδιάγραμματα της όλης διαδικασίας ώστε να μπορούμε να βρούμε τις σωστές χρονικές στιγμές και να έχουμε υπόψη μας τους χρονικούς περιορισμούς όσον αφορά την προτινόμενη εξαίρεση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προτείναμε αναβολή ενός έτους. Έτσι διατηρείται η μόχλευση και αφαιρείται οποιαδήποτε δικαιολογία από τους εταίρους τρίτων χωρών που διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει τις δικές τους διαδικασίες ε, στο πλαίσιο της ΕΚΑΟ και δεν μπορεί να ε, παρέχει ένα αποτέλεσμα σωστό υλοποιώντα μια τέτοια διαδικασία, ενώ η διαδικασία προετοιμάζεται για τη συνέλευση. Αυτή η δυναμική έχει πάψει να υπάρχει. Αυτό που έχουμε τώρα είναι μια πραγματική αυθεντική ευκαιρία συμμετοχής όλων των εταίρων και δέσμευσής τους. Και πραγματικά εμείς προσδοκούμε ότι οι εταίροι από τρίτες χώρες θα απαντήσουν θετικά κυκλοφόρησαν κάποιες εκθέσεις και κάποιες φήμες που λένε ότι οι υπαδιστάζουν για ένα ενιαίο μέτρο. Θα πρέπει να συζητήσουμε με όλους αυτούς τους εταίρους, να τους παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και αυτό έχει ήδη γίνει πριν από το, συνάντηση του Συμβουλίου του ΙΚΑΟ τον Νοέμβριο. Πιστεύω ότι έχουμε σταθερά θεμέλια για να συνεχίσουμε αυτό τον διάλογο μέσω διαδικασίες υψηλού πολιτικού επίπεδου αλλά και μέσω διμερών ανταλλαγών μεταξύ εμάς και των τρίτων χωρών, των εταίρων μας σε τρίτες χώρε, που ίσως δεν έχουν καταλάβει τις προθέσεις και τις συνέπειες του ETS της Ευρώπης. Η εξοεδαφική πτυχή κατά την άποψή μα θα επιτρέψει να υπάρξει περιθώριο για ένα ε, ικανοποιητικό αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο από την ΙΚΑΟ. Μετά από την υιοθέτηση από τους επιτρόπους στις 20 Νοεμβρίου της πρότασής μας ε, είχαμε ήδη τις συζητήσεις ομάδα εργασίας για αυτό το θέμα. Οι επόμενες συζητήσεις έχουν προγραμματιστεί στις 7 Ιανουαρίου. Πολύ σύντομα δηλαδή τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν πλήρως. Και τα σχόλια που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής ε, δεν ε, δεν εναντιώνονται ριζικά στην πρόθεση και στη λογική της πρότασης. Πιστεύω ότι συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει αυτή τη θέση. Ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική, πιστευτή, αξιόπιστη γραμμή όσον αφορά την υλοποίηση της πρότασής μας. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι και οι διαπραγματευτές μας στον ΙΚΑΟ θα έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας όσον αφορά την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων σε ένα μέσο ενός διεθνούς καθεστώτος, της εφαρμογής ενός διεθνούς καθεστώτος. Εμείς ως Κομισιόν είμαστε ιδιαίτερα διατεθειμένοι να προβούμε σε συζητήσεις, να εξηγήσουμε αυτή την πρόταση σε οποιοδήποτε μέλος ε, του προσωπικού του Κοινοβουλίου ενδιαφέρεται. Και θα δώσουμε πληροφορίες το συντομότερο δυνατό για τα διάφορα στάδια. Ήδη online, έχουμε ε, δημοσίευση υλικό συχνών ερωτήσεων όπου εξήγεται ποιες χώρες θα καλύπτονται, ποιο είναι το υλικό, ποιες είναι οι συνέπειες της υλοποίησης, της νομοθεσίας και της σχετικής πρότασης. Καλώ τους συναδέλφους να διαβάσουν αυτό το υλικό και θα προσθέσουμε και άλλες ερωτήσεις και αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις ευχαριστώ θα τις απαντήσουμε μέσω της Γενικής Διεύθυνσης ε, Climate. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Και τώρα ο εισηγητής Πέτρα Λίζα για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί προχώρησε πάρα πολύ ο χρόνος. Το θέμα των εθνικών τελών αναφέρθηκε από συνάδελφο. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να το δουν αυτό. Έχουμε ένα έγγραφο που έχει διανεμηθεί. Αν κάτι δεν πάει καλά, να μου το αναφέρετε γραπτός. Αμέσως ε, θα ζητήσουμε να υπάρξει επανόρθωση. Η διάσταση όμως, η κατεύθυνση είναι σαφής. Απευθύνομαι και στους Βρετανούς συναδέφους και στους συναδέφους ε, των συντηρητικών, των Tories, ε, σε σχέση με την έγκριση της έκθεσης που τότε ανήκαν στο ΕΛΚ. Η Βρετανική κυβέρνηση πρόσφατα, υπό την ηγεσία των Tories και των φιλελεύθερων, αύξησαν τα τέλη για τις εναερίες μεταφορές. Όταν ταξιδεύει κανείς με πρώτη κατηγορία, σε, στην πρώτη κατηγορία, ισχύει αυτό, αλλά πληρώνουν και για στην την οικονομική θέση. Και να δώσω ένα ακραίο παράδειγμα. Αν έχουμε 6.000 μίλια διαδρομή, για παράδειγμα, από το Λονδίνο στην Ασία, 184 λίβρες ανά άτομο, εντάξει, στο μεταφορικό έργο ένα ενιαίο τέλος σε ένα κράτος μέλος. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων και να λειτουργεί αυτό όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα χρόνο στην Ευρώπη να περιοριστεί και στις διπηρετικές να συμπεριληφθεί μετά από ένα έτος ή να ξεκινήσει μια παγκοσμιοποιημένη προσέγγιση θα δημιουργηθεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Αν αυτά τα 184 ή 184 λίμπρες ισχύουν έτσι είναι πολύ μετριοπαθής ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα θα υπάρξει, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη των ε, ταξιδιωτών μέχρι ότου να υπάρξει τελική πτώση. Δεν γίνεται αυτό. Λόγω της αύξησης λέει των ε, κομίστρων, λόγω των, της εμπορίας ρήπων. 25 είναι αυτό πράγματι ε, τόσο ε, επιβαρυντικό. Αναφέρθηκε από τον πρόεδρο, αναφέρθηκε το παράδειγμα των ανατολικών φρισλανδικών νησιών. Όταν ο πρόεδρος ε, θέλει να κινηθεί στη δική του εκλογική περιφέρεια ή ένα μέλος της εκλογικής του περιφέρειας από την πατρίδα του θέλει να πάει στην περιφερειακή πρωτεύουσα, πληρώνει το δεκαπλάσιο. Δεν γίνεται αυτό να κάνουμε λόγο δηλαδή με αυτόν τον τρόπο για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσω των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν τα κράτη-μέλη βάζουν το χέρι στην τσέπη των πολιτών ανέσχυντα με αυτόν τον τρόπο. Το δέχεται ο τύπος, το δέχονται οι εταιρείε εναέριων μεταφορών, το δέχονται όλοι και ασκούν πίεση και επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκείνοι το κάνουν αυτό επειδή πιστεύουν ότι είναι αποδυναμωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με αυτήν. Είμαι πρόθυμος να συζητήσω οποιαδήποτε πρόταση και να εξειδικεύσουμε και τις διατυπώσεις. Να δουλέψουμε γοργά ώστε να εκπονηθούν οι τροπολογίες. Να έχουμε αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο έκθεσης που θα προτείνουμε ώστε να έχουμε τη δυνατότητα όλες οι προτάσεις, όλες οι τροπολογίες να ενταχθούν έγκαιρα στο σωστό πλαίσιο. Δούλεψε πολύ προσεκτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να κινηθούμε. Πολλά πράγματα που αναφέρονται στη συζήτηση σταθμίστηκαν προηγούμενα, αξιολογήθηκαν. Γι' αυτό δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τόσο σημαντικά αυτή την πρόταση. Σε ένα σημείο μια επισήμανση, μια αποσαφήνιση απαιτείται. Διευκρίνηση, επειδή ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπα και εγώ, δεν θα έχουμε παγκόσμια συμφωνία που από την 1η του 2014 να αρχίσει να ισχύει. Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε όμως από την ΑΙΚΑΟ όχι να έχουμε μόνο ένα πλαίσιο για τις περιφερειακές και εθνικές εκπομπές ρήπων, αλλά ε, μια σαφή δέσμευση στην οποία θα μπορούμε να βασιστούμε αξιόπιστα ότι κάποτε θα καταλήξουν σε μια παγκοσμιοποιημένη λύση και αυτό είναι όρος και προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει πρέπει να ισχύει, να ασκηθεί πίεση ώστε αυτά τα οποία προτείνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο ερωτήσεις απαντήσεις, questions and answers, μια παγκοσμιοποιημένη συμφωνία να είναι ο στόχος. Και τώρα χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο, επειδή όλα αυτά δεν μπορούν πρόθεσμα να επιτευχθούν. Ένα πλαίσιο που εμείς και άλλοι να μπορούμε να ρυθμίζουμε το δικό μας περιφερειακό σύστημα πτήσεων προσαρμοσμένο όπως απαιτείται. Δεν γίνεται μέχρι το 2020 το 2025 να μην κάνουμε και τίποτα, να σταυρώσουμε τα χέρια. Δεν θα ήταν ικανοποιητική αυτή η λύση με κανένα τρόπο. Ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάναμε. Είμαι πρόθυμος να δεχθώ προτάσεις σας με τροπολογίες σας. Είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, πιεστικό. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και παρόλα αυτά την άνοιξη του 2013 να ολοκληρώσουμε. Να στείλουμε, να σηματοδοτήσουμε με σαφήνεια ότι αν υπάρχει προοπτική για μια διεθνή συμφωνία δεν θα κολλησιεργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και θα συνεργαστούμε να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Θα καταβάλουμε τη δική μας συνεισφορά. Ευχαριστώ. Αγνόησα τη συνάδελφο Φώστερ που έχει ζητήσει τον λόγο. Έχετε τον λόγο πάρα. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση στην οποία δεν απήντησε η Κομισιόν. Πολλοί είπαν ότι ισχύει αυτή η εξαίρεση για 12 μήνες. Δεν, δεν λέω, ξέρω τι ποιο είναι το πρόβλημα με τη Lufthansa και αυτά μιλάμε και για τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Εν πάση περιπτώσει, 12 μήνες είναι η ισχύ και εάν δεν ε, γίνει τίποτα μετά τα, τους 12 μήνες, άσχετο ότι θα κάνει η ΚΑΟ, θα υπάρξουν κυρώσεις προς τις μεταφορείς τρίτων χωρών θα υπάρξουν κυρώσεις, γιατί ξέρετε ότι δεν θα συμμορφωθούν οι <coughs> μεταφορείς τρίτων χωρών. Εγώ ξέρω, είμαι βεβαία ότι στο πέρας των 12 μηνών δεν θα ε, ε, συμμορφωθούν οι αερομεταφορείς των τρίτων χωρών. Τότε θα υπάρξουν κυρώσεις. Κυρία Φώστερ, νομίζω ο σωστό εταίρο ε, είμαστε εμεί. Εμεί αποφασίζουμε αυτό, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα για να υποβάλει πρόταση. Εμεί θα αποφασίσουμε ω Ευρωβουλή τι θα γίνει στο τέλο τέλο, τι θα ενταχθεί στην έκθεση του Πέτερ Λίζε και τι θα καταλήξει εκεί. Αν θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Εγώ ως νομοθέτης θεωρώ ότι είναι το έργο μας, δικό μας έργο, όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Μπορώ να απαντήσω την ερώτηση. Ο νόμος θα εφαρμοστεί σε όλους τους αερομεταφορείς που ε, ε, κάνουν εσωτερικά δρομολόγια, διευρωπαϊκά δρομολόγια, ασχέτως εθνικότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κυρώσεις ε, υπό την Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Ναι, το σχέδιο έκθεσης ε, θα το εξετάσουμε στις 23 Ιανουαρίου, θα το συζητήσουμε. 28 Ιανουαρίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 18 Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, προς έγκριση. Θα έχουμε την ψήφιση τελικά στην Επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου 2013 και το σύνολο θα καταλήξει, ελπίζουμε, το Μάρτιο στην Ολομέλεια προς έγκριση. Και έτσι λοιπόν η συζήτηση εδώ ολοκληρώθηκε επ' αυτού. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη εδώ. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για την γνωμοδότηση 2011 για την απαλλαγή 2011 και διάφορα θέματα δεν θα σας τα διαβάσω. Όλα θα μας τα πει Γιούτα Χάουκ, το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, που είναι εδώ η εισηγήτρια για αυτά. Παρακαλώ Γιούτα Χάουκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω λοιπόν ταχύτατα τα σημεία, επτά σημεία τα οποία καλύπτονται, γιατί είναι 7, ενημερωτικά, Utah Hawk. Πρέπει τώρα, όχι ταχύτατα, έχουμε χρόνο μέχρι τις 7. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν χρειάζεται να τα πας ε, ε τι, ως λέλαπα. Εντάξει, ναι, αλλά έχουμε και άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη που πρέπει να καλύψουμε. Εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε και από αυτό, αν έχουμε, σε σχέση με την λήψη απόφασης, την ε, απαρτία ή την ικανότητα λήψης απόφασης, δεν χρειάζεται βέβαια να ληφθεί απόφαση, αν δεν έχουμε απαρτία θα μπορούσαμε να πούμε. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό 2011 και για την χωρίση απαλλαγή. Δεν θέλω τώρα εδώ να μακρηγορήσω με κανένα τρόπο. Απλά και μόνο να πω τούτο. Γενικά για τις, ε, τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες, στη δική μας ε, ευθύνη εμπίπτουν πέντε από αυτούς τους οργανισμούς. Και γενικά τώρα για αυτά Έχουμε και μια άλλη έκθεση όπου κάποιες αρχές αναφέρονται και περιγράφονται. Τώρα πρέπει να υπενθυμίζουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάποιες αρχές δημοσιονομικές που η ίδια η συνθήκη και ο ίδιος ο κανονισμός μας, ε, μας δίνουν και πρέπει να τηρούνται αυτές οι αρχές. Τήρηση και ενιαίο πλαίσιο προϋπολογισμού. Σε αιτήσια μορφή η υποβολή του προϋπολογισμού και η αντιστάθμιση και ο ισοσκελισμός. Οι συνάδελφοι που θα έχουν κάπως λίγο προσέξει κατά την τελευταία εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου θα γνωρίζουν ότι το Συμβούλιο, τουλάχιστον εκείνο το οποίο ε, πρέπει να λάβει, λαμβάνει υπόψη, είναι ο ισοσκελισμός. Για τον προϋπολογισμό 2013, 9 δις ευρώ αναλαμβάνονται ως χρέη. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ με τον ισοσκελισμό. Αυτό είναι παρόδο, εν πάση περιπτώσει. Είπα για άλλη μια φορά ότι ο ετήσιος χαρακτήρας δημοσιονομικά πρέπει να ισχύει για όλους και για τους οργανισμούς. Ετήσιος χαρακτήρας τι σημαίνει. Τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται δεν μπορούν απλά και μόνο να κινούνται και να μεταφέρονται μέχρι το επόμενο έτος δημοσιονομικά. Πρέπει ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός να, γίνονται, να γίνεται με τέτοιο καλό τρόπο, με τακτά πλαίσια και διαδικασίες, ώστε να διατίθενται αυτά τα κονδύλια, να καταβάλλονται όπως προβλέπεται. Αν εξαίρεση. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται, απαιτείται διαφάνεια. Χρειάζονται πληροφορίε γιατί συνέβη αυτό και δεν αντλήθηκαν αυτά τα κονδύλια, δεν καταβλήθηκαν τα ποσά. Αν δείτε τι προτάσει μου για τη γνωμοδότηση αυτή, τι λέμε. Σε, κάποιες, σε κάποιους οργανισμούς πάλι απαριθμούνται ότι απαριθμούνται τα στοιχεία για τα οποία οι οργανισμοί αυτοί είχαν κάποια προβλήματα, κάποιες δυσκολίες τα δεσμευμένα αυτά ποσά, τις πιστώσεις υποχρεώσεων που δεν μπόρεσαν να τι ε, καταβάλουν, να τι εκτελέσουν με κάποιε συμβάσει που είχαν. Δηλαδή, οι πληρωμέ μετατίθενται για το επόμενο δημοσιονομικό έτος. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα σχετικά. Λέμε όμω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται, εκπροσωπείται σε όλα τα συμβούλια όλων αυτών των οργανισμών, σε όλα τα εκτελεστικά συμβούλια, πρέπει ως αρρωγός να ανακουφίσει την κατάσταση κατάσταση, να συνδράμει τους οργανισμούς. Δηλαδή και το σημερινό προγραμματισμό όπως ε, έχει, ε, έχουμε καταλήξει αλλά και για τις ε, προκηρύξεις για τη στελέχωση με προσωπικό αυτών των οργανισμών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με common approach, με κοινή προσέγγιση, συζητήσαμε επί τρία χρόνια για αυτά τα θέματα και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι σκέπτεται να κάνει και πώς μπορεί να συνδράμει αυτούς τους οργανισμούς έχει σαφείς ενδείξεις. Πρέπει όμως να πούμε ότι το κάναμε αυτό και στο παρελθόν πριν από το Common Approach. Είχαμε καταφέρει να περάσουμε να έχουν ε, σχέδια και προγράμματα δεσμευτικού χαρακτήρα για τη στελέχωση και το προσωπικό τους. Πρέπει να πούμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εταίροι γενικές διευθύνσεις πρέπει να προσέξουν σε τέτοιες περιπτώσεις όταν μετατίθενται κονδύλια να ασκούν πίεση να τηρούνται τα προγράμματα και οι σχεδιασμοί. Δεν μπορεί να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ριζοσπαστικά άρδιν εκβάθρον να αλλάζει την, ε, τα προγράμματα στελέχωσης αυτών των οργανισμών με τον Ιστέρη. Πρέπει μια στιγμή να πιω κάτι γιατί βράχνιασα, συγγνώμη. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είχα να πω και τώρα ουσιαστικά αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε για τους οργανισμούς αυτή η παρατήρηση δύο άλλα ακόμα στοιχεία πρώτον και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι ας το πω έτσι ε, ο, ο, ο τελευταίος ας το πω έτσι ε, κριτής ε, θεσμικών οργάνων και αυτό εργάζεται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε ένα χρονοπλαίσιο. Και αυτό που βλέπουμε με την έκτακτη έκθεση που συνέταξε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων ή αρμοδιοτήτων μέσα σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή οργανισμό και πάλι η φθορά του χρόνου πρέπει να δούμε ότι έχει, έχει προχωρήσει ε, δεν έχουν παραμείνει οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί στο σημείο το οποίο έλεγξε κάποτε το ελεγκτικό συνέδριο, τα πράγματα προχώρησαν, μετεξελίχθηκαν. Υπάρχει μια ανέλυξη και έχουν εκπονήσει μηχανισμούς και έχουν μετεξελιχθεί και έχουν προσαρμοστεί σε σχέση με την επίλυση ή αντιμετώπιση των διαφορετικών καταστάσεων συγκρούσεων συμφερόντων ή προς αποφυγή αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων. Αυτό που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι απόλυτα επικαιροποιημένο, δηλαδή δεν είναι απόλυτα ενημερωμένο. Δεν αποκρίνεται στην κατάσταση πραγμάτων κατά τα τέλη του 2012 ή κατά την έναρξη του 2013. Και ένα ακόμα επιπλέον σημείο. Τώρα, για, για την ε, υπηρεσία για τα φάρμακα για την, την ιατρική υπηρεσία. Είπαμε και λέγαμε πάντα ότι παρακαλούμε πρέπει να εργάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται τα κόστη τους, οι δαπάνες τους. Για την κάλυψη των δαπανών πρέπει να εισπράττουν έσοδα τα οποία θα αντισταθμίζουν και θα ισοσκελίζουν τις δαπάνες τους. Για την τάξη όμως πραγμάτων των εσόδων τους δεν είμαστε δόξα το Θεό εμείς οι νομοθέτες, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο. Τι κάνει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Συναπαρτίζεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών που αποστέλλονται εκεί και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για να καλύπτουν τα έσοδά τους στις δαπάνες διότι τα κράτη-μέλη α uh, με τις εισφορές τους εμπλέκονται. Εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους πούμε σας παρακαλούμε να δημιουργήσετε μια νέα τάξη εσόδων, ένα νέο κανονισμό εσόδων, να ισοσκελίζονται τα έξοδά σας. Να δούμε τι θα κάνουν λοιπόν τώρα επιτέλους. Αυτές οι παρατηρήσεις για τους οργανισμούς. Τώρα με δύο λόγια αγοργά να έρθω στο σημείο το επόμενο της ημερήσιας διάταξης, το οποίο ως οκτώ στη σειρά, όχι οργανισμοί, αλλά τμήμα 3. Γενικός προπολογισμό, γενικός προϋπολογισμός της Επιτροπής. Τμήμα 3. Λοιπόν και πάλι πρέπει να καταλήξω στο να πω ότι προσέξτε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δουλεύει απόλυτα ορθά και σωστά. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει με κάποια κακεντρέχεια ότι είναι μάλιστα μεροληπτή. Γιατί? Γιατί τι έκανε. Παρουσίασε απλά στην ετήσια έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο και είπε οι τομείς πολιτικής ε, περιβάλλον και υγείας αποκινούμε την ανάπτυξη της υπαίθρου και την αλληλεία παρουσιάζονται και διαφωτίζονται. Πράγμα το οποίο έχει σαν ε, επίπτωση να γίνεται αμέσως λόγος για το ποσοστό σφάλματος. Σφάλματος 0,25% πόσο είναι. Δεν μπορώ να το πω τώρα ακριβώς ποιο διαπιστώνω ότι είναι. Αυτά όμως τα οποία εντάσσονται στη δική μας αρμοδιότητα, δηλαδή περιβάλλον και υγεία, δεν έχουν, καμιάς, δεν έχουν κανένα ποσοστό σφάλματος. Μηδενικό σφάλμα. Και δεν είναι εντάξει λοιπόν όταν αυτά τα ρίχνουν σε ένα σακί με άλλες υποθέσεις όπου υπάρχει ποσοστό σφάλματος. Στην επόμενη έκθεση λοιπόν, στην χωρίση απαλλαγή 2012 πρέπει με διαφορετικό τρόπο να παρουσιαστούν τα πράγματα. Διότι διαφορετικά μια στρεβλωμένη εικόνα, εικόνα απόλυτα στρεβλωμένη εικόνα περνάει προς τα έξω για την υγεία και το περιβάλλον. Δηλαδή, για την ικανοποίηση για το πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα ε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές, η Γενική Διεύθυνση για τα θέματα κλίματος, ε, μια νέα Γενική Διεύθυνση με φιλόδοξο, α το πω έτσι, χρονοπλαίσιο του έργου, είναι σαφές, ε, το κατανοούμε, αυτό το οποίο γίνεται είναι όλα υπερβολικά αισιόδοξα ίσως τα οποία είχαν ε, ε, αρχικά συλληφθεί. Έχουμε ένα ποσοστό 58% ποσοστό εκτέλεσης. στη συνέχεια θα αλλάξουν τα πράγματα. Όταν θα έχουμε τη χορήγηση απαλλαγής 2012 θα έχουν τα πράγματα αλλάξει και δεν θα είναι όπως είναι σήμερα. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα σε όλα αυτά. Για όλους τους οργανισμούς, για όλους τους οργανισμούς και οργανώ, υπηρεσίες και για την ε, Επιτροπή συνιστώ το εξής, να χορηγηθεί απαλλαγή, να υπερψηφίσετε τη χορήγηση απαλλαγής. Γιούτα Χάουξ, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η σύστασή σου, χορήγηση απαλλαγή, υπεψήφισή τη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Κανένα δεν μπορεί τόσο ζωντανά να παρουσιάσει αυτά τα α το πω έτσι ανούσια και βαρετά στοιχεία όπω η γιούτα Χάουκ τα οποία τα ζωογονεί η ίδια με τη ζωντανή παρατήρηση, παρουσίαση. Και, και στη συνέχεια Βέρλιν και εγώ. Ναι, συγγνώμη, δεν είδα συνάδελφε, Σκιώδη εισηγητής, εσείς έχετε τον λόγο πρώτα, παρακαλώ σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους και ιδιαίτερα την Γιούτα Χάουγκ που για άλλη μια φορά έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ. Θα είμαι πολύ γοργός και δεν θα επαναλάβω, δεν θα όλα αυτά τα οποία είπε η Γιούτα Χάουγκ όσον αφορά τις παρατηρήσεις συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτέ. Ένα σημείο όμω θα ήθελα να αναφέρω στη συζήτηση και αυτό είναι η σκοπιμότητα της σύνταξης της έκθεσης, του τρόπου που έχει η έκθεση και η διατύπωσή της και που θα προτιμούσα να ήταν κάπως διαφορετική. Σε, όλες, σε όλους τους οργανισμούς εμφανίζεται μια διατύπωση, μια φράση αυτού του είδους σχεδόν ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο οργανισμός εκτέλεσε τον ε, προϋπολογισμό με αντίθετο τρόπο από την αρχή του κόστους οφέλους. Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για απάτες ή παρατυπίες Φαίνεται ότι λέγοντας αυτό υπήρχε κάποια προϋπόθεση ότι θα ήταν λέει ομαλό να υπάρχει παρατυπία, απάτη, να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ή σε σχέση με τις αποδείξεις για την αρχή της αποτελεσματικότητας των δαπανών, δηλαδή την αλλαλογικότητα του, των δαπανών ως προς το όφελος. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε λέει αποδείξεις ε, για κάτι τέτοιο, ότι να συμβαίνουν παρατυπίες ή απάτες. Θα έλεγα ότι καλύτερο θα ήταν να μην είχαμε μια τέτοια φράση. Να μην διατυπώναμε αυτό το πράγμα με αυτή τη διατύπωση. Να είχαμε μια διαφορετικού τύπου διατύπωση που απλά να έλεγε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούμε να χορηγήσουμε την απαλλαγή και τα πράγματα βαίνουν καλώς. Και εντάξει, να χορηγήσουμε αυτές τις απαλλαγέ που αναφέρθηκαν προηγούμενα από την κυρία Χάουγκ. Όμως, ο κοινό τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται αυτά πολλές φορές και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι αναφορές π.χ. από το ελεγκτικό συνέδριο υπάρχει μετέωρη, μια υποψία ή μια ίσως ενδυνάμει καταγγελία ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιες απάτες ή τέτοιες καταχρήσεις ή παρατυπίες, αλλά δεν βρήκαμε αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Εφόσον λοιπόν δεν βρέθηκαν τέτοιες αποδείξεις και τέτοια τεκμήρια, και σε σχέση με την αναλογικότητα ωφέλους και αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις δαπάνες υποθέτουμε ότι οι αρχές της χρηστής διαχείρισης, διακυβέρνησης της οικονομίας και η αρχή της αποτελεσματικότητας ισχύουν και έτσι πρέπει να ακολουθηθούν. Πρέπει όμως αυτό να λέμε ότι ή βαίνει καλός κάτι ή όχι. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια που χρησιμοποίησε με τον τρόπο αυτό αυτή την ε, αναφορά και αυτό το σημείο με αυτόν τον τρόπο ε, αναφέρεται για τη χορήγηση απαλλαγή στους οργανισμούς με τον τρόπο που ανέφερε. Ευχαριστώ. Φανώνει παρακαλώ. Στη συνέχεια έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην κυρία ΣΥγητρια για την ποιότητα των κριτήριων που έχει περιλάβει. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα αυτής της ετήσιας συνάντησης. Η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό δημοκρατικού ελέγχου, όπως ε, προσδοκείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη συνθήκη, παραχωρεί την απαλλαγή στην Κομισιόν όχι μόνο αφού έχει επιβεβαιώσει την νομιμότητα και την ορθότητα των λογαριασμών, αλλά και αφού έχει υπηλθεύσει την ποιότητα των δαπανών ως εκπρόσωποι των πολιτών θεωρούμε ότι κύριο καθήκον μας είναι να αξιολογήσουμε φυσικά για τις πολιτικές δημοσίες υγείας, περιβαλλοντός και ασφάλειας των τροφίμων κατά πόσο οι πέντε οργανισμοί που υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές έχουν δαπανίσει τους φόρους των φορολογουμένων σωστά. Κατά πόσο δηλαδή αυτά τα κονδύλια έχουν επιτύχει πραγματικά τους πολιτικούς στόχους για τους οποίους έχουν διατεθεί η ασφάλεια των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε, ο έλεγχος και η διαχείριση των ασθενειών, η ποιότητα των τροφίμων που τρώμε, η υγεία, η καθαρότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε είναι θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας. Έτσι λοιπόν αυτή η διαδικασία απαλλαγής ε, ειδικότερα σε αυτή την περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης όπου δυστυχώς ε, φαίνεται να τροφοδοτείται σημαντικό αντιευρωπαϊκό συνέστημα όπου πολλοί πολίτες λένε ποια είναι η Ευρώπη να μας ζητάει να κάνουμε σημαντικές θυσίες για την υποστήριξη σημαντικών προπολογισμών. Εδώ πρέπει να υποστηρίξουμε τους πολίτες μας και να τους πούμε ότι τα κονδύλια που έχουν αφιερωθεί σε στρατηγικά μέσα της, μέσα, της Επιτροπής μας είναι αιτιολογημένες είναι αιτιολογημένα αυτά τα κονδύλια και ότι βοηθούν να προσφέρεται τη θεμενή αξία και ότι αποφεύγονται τα περιτά έξοδα. Για να στείλουμε αυτό το μήνυμα πρέπει οπωσδήποτε σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγής να ε, δείξουμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα και να αξιολογήσουμε κατά πόσο μετά από ένα χρόνο έχουν αξιοποιηθεί οι συστάσεις, έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις του προηγουμένου έτους, έχουν ληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες βελτίωσης της κατάστασης των πραγμάτων. Όπως γνωρίζετε, όσον αφορά γενικότερα τους διάφορους οργανισμούς, όπως και τους δικούς μας πέντε οργανισμούς που εμπίπτουν στη δική μας αρμοδιότητα, συναντάμε πάντα τα ίδια προβλήματα. Την έλλειψη αποτελεσματικών διαδικασιών για την καταπολέμηση τυχών διενέξεων συμφερόντων που όπως γνωρίζουμε πέρυσι το περσινό έτος ε, ε, αφορούσαν την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Τροφίμων αλλά και τη διαχείριση ε, ανθρωπίνων πόρων για πιο διαφανείς διαδικασίες και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Όπως ε, τονίζει η συγγητριά μας, φαίνεται ότι το 2011 επιτεύχθηκαν σημαντικές πρόοδοι, τουλάχιστον όσον αφορά τον Οργανισμό Περιβάλλοντος και τον Οργανισμό Ασφαλής των Φαρμάκων. Το ελεγκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του διαπίστωσε κάποια λάθη σε πληρωμές για το περιβάλλον, τη γεωργία και την αλία, αλλά ταυτόχρονα όπως υπογράμμισε η συγγήτρια στο σύνολο τα ποσοστά εκτέλεσης συνολικά των κονδυλίων του προπολογισμού σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής μας είναι ικανοποιητικά. Χάρη σε αυτές τις διαπιστώσεις και δεδομένου ότι Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων δεν φαίνεται να υπάρχουν απάτες ή σημαντικά σφάλματα. Η εισηγήτρια πολύ σωστά συνέστησε να εκχωρήσουμε την απαλλαγή στις πέντε επιτροπές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας. Θεωρώ εγώ ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε από τη δική μου πολιτική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση η ορθότητα και η νομιμότητα των λογαριασμών αυτών των οργανισμών θα υφιστούν θα υποστεί ούτως ή άλλως σε περαιτέρω πιο συγκεκριμένη βάθυνση από τον συνάδελφο Μπέρμαντι, τον οποίο εκτιμάμε και εμπιστευόμαστε ιδιαίτερα στην Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. τελευταία αλλά σημαντική παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ θαυμάζω ιδιαιτέρως την ε, Ρώμη, το σθένος της ε, εισηγητρίας που θαύμασα άλλωστε και στους πρόσφατους τριμερείς ε, διαλόγους για το 2020. Θα πω πώς βλέπει η ομάδα μου τις απαλλαγές. Εμείς δεν δίνουμε τις ε, απαλλαγές από τη στιγμή που ε, δεν ε, έχει δοθεί πράσινο φως για τον προϋπολογισμό από τους ε, OECD guidelines and in order to ensure the highest quality of internationally recognized. Από το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, και ε, επομένως θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να δώσουμε απαλλαγή στα επιμέρους τμήματα. Ε, θα πω και δύο λόγια. Θεωρούμε ότι είναι μια καλή στιγμή, μια καλή ευκαιρία αυτή η συζήτηση για τις απαλλαγές γιατί δείχνει ότι συνήθως έχουμε προβλήματα αλλά τελικά ε, τα ξεπερνάμε. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας αυτή τη φορά να είμαι πιο στεναρή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην, ε, ε, την παρατήρηση της Μαρίνας Γιανακουδάκη, της συναδέλφου μου, της συναδέλφου Ε, γιατί στην παρατήρηση της ε, σχετικά έλαβε την απάντηση ότι θα, υπήρξαν, θα υπήρχαν μάλλον πιο ε, σωστές αντιμετωπίσεις των επιμέρους προϋπολογισμών και ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία ε, αναθεώρησης και ε, ε, ε είχε πει κιόλα ο υπεύθυνο του Συμβουλίου ότι ε, θα τις έδινε τα απαραίτητα εχέγγυα, εχέγγυα τα οποία εγώ δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή εδώ και επομένως δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση απέναντι στη διαδικασία. Επομένως, επομένως για μία ακόμα φορά δεν θα υπερψηφίσουμε ε, την απαλλαγή, απλώς συμμετέχουμε στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα. Πρωτού δώσω τον λόγο στον εισηγητή, θα δώσω τον λόγο στην Επιτροπή, παρακαλώ, εσείς. Okay, next Okay, dann die Kommission hat sich nicht geeinigt, dann gebe ich der Berichterstatterin. Δίνω τον λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια, εφόσον δεν παρέμβει η Επιτροπή. Λοιπόν, για να το πω, είναι ακριβώς αυτό το δίλημα. Σοβαρά τώρα, το δίλημα. Και μάλιστα όχι μόνο σε σχέση με τη, τα τμήματα της Επιτροπής, αλλά και τους οργανισμούς. Δηλαδή, οι οργανισμοί απλά δεν μπορούν να βασιστούν στις ε, εταίρους που έχουν γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε καν όταν πρόκειται για την κατάρτιση του προϋπολογισμού σχεδίου. Και θα έλεγα, αυτό είναι η κατάδειξη ανάγλυφα αυτών που πάντα λέγαμε και λέμε. Ότι δηλαδή μια κανονική η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει τουλάχιστον να έχει αρκετή γνώση για τον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά και τους συσχετισμούς των θεμάτων ώστε οι αρμόδιοι να μπορούν να λογοδοτήσουν και να δώσουν λογαριασμό και απαντήσεις. Δεν, απαντώ τώρα, δεν απαιτώ να προσέρχονται στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά να ξέρουν περί τίνο πρόκειται και να είναι αυτά τα οποία λένε αξιόπιστα και βάσιμα. Τώρα, για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, στην Τζούντι, να πω τούτο αυτό με τη μη χορήγηση απαλλαγής που είπες δεν το κατάλαβα απόλυτα. Διότι είπε, ίσως ε, είναι θέμα διατύπωσης ή διερμηνίας ε, που θα ήθελα εδώ να, το, να διαφοροποιηθούμε από αυτού. Είπε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει λέει ολοκληρώσει ακόμα το οικονομικό έτος όμως 2011 έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και τι έκανε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τους οργανισμούς, τι είπε, έδωσε πιστοποίηση σε όλους τους οργανισμούς ότι και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά και ίσως υπάρξει κάποια τροπολογία του Ζωζέ Μανουέλ δεν βρέθηκαν λέει παρατυπίες δεν ανακαλύφθηκαν παρατυπίες και όλα έβαιναν καλώς και έβαιναν εν τάξη. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, αν η Τζούντι το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο το απαιτεί να ισχύει για όλους τους οργανισμούς, δεν ξέρω ακριβώς τι φαντάζεται υπό αυτή τη διατύπωση, αλλά μόλις το είπα. Υπάρχει αυτή η common approach, όπως την αποκαλούμε. Με άλλα λόγια, τι έχουμε. Σε πολλές και αλλεπάλληλες συνεδριάσεις τι κάναμε. Και το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήλθαμε και εκπονήσαμε και αποφασίσαμε, εγκρίναμε αυτή την κοινή προσέγγιση, common approach. Από την ε, μία πλευρά ήταν ο Giles Chichester σε αυτή την ομάδα εργασίας μέλος που είχε ε, ασχοληθεί με αυτό. Και γι' αυτό τώρα, πέρα από το ότι αυτό το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι στη διάθεση όλων και υπό τη Δανέζικη Προεδρία ήδη το εγκρίναμε και ο πρόεδρος, ο δικός μας πρόεδρος, το προσυπέγραψε και ο πρόεδρος της ε, ε, Προεδρίας του Συμβουλίου της Δανίας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο αντιπρόεδρος, δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς ποιος ήταν. Εν πάση περιπτώσει, προς τον κύριο Σανώνη θα ήθελα να πω το εξής. Και πάλι με τη δική σας παρατήρηση δεν είμαι βέβαιος αν έγινε κάποιο σφάλμα ή κάποια παρερμηνία από τη γλώσσα αυτή. Δεν καταλαβαίνω Ιταλική βέβαια το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ακούστε, δεν ούτε ένα σφάλμα δεν διαπίστωσε. Ούτε για το περιβάλλον, ούτε για το, τον τομέα υγείας. Μόνο αυτό που έκανε τι ήτανε. Πήρε το περιβάλλον και πήρε και τον τομέα της υγείας και τα ε, ε, ε, ενέταξε με την πολιτική για την αλληλεία και για την πολιτική με την ανάπτυξη υπαίθρου σε ένα συνονθήλευμα και είπε ποσοστό σφάλματος 5,2% ενέχεται εκεί. Όμως περιβάλλον και υγεία δεν έχουν κανένα λάθος ποσοστό σφάλματος, μηδενικό ποσοστό σφάλματος. Αλληλεία και ανάπτυξη υπαίθρου είχαν ποσοστά σφάλματος. Και έτσι ίσως απορρέει η ιδέα ότι και το ε, ποσοστό σφάλματος καλύπτει την υγεία και το περιβάλλον. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Δεν συμβαίνει. Και θα έπρεπε να υπήρχαν και εδώ εκπρόσωποι που θα το αποσαφήνιζαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Απαιτώ από το ελεγκτικό συνέδριο να επιλέξει μια άλλη μορφή παρουσίασης των πραγμάτων, ώστε να είναι σαφή και διαφανή αυτά τα οποία λένε Ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Για το 0,76% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο το θεωρούν γελίο υπερβολικά μικρό ποσοστό και δεν θέλουν να αφιερώσουν μια πρόσθετη αράδα, μια γραμμή για ένα τέτοιο θέμα. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να γίνει και να αποσαφινιστούν τα πράγματα διότι μπορεί κανείς να αποκομίσει λάθος εντύπωση από αυτή την παρουσίαση. Πρόεδρε, <clears throat> για την ε, την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια για να είναι σαφή τα πράγματα σχετικά. Πρόεδρος, ναι, αμέσως θα το κάνουμε αυτό. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο θα παρέμβει για λογαριασμό τη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δίστασα λίγο διότι δεν είχα φανταστεί ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ερωτήσεις για την Κομισιόν στις διάφορα σχόλια που ακούσαμε. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι ωφέλιμο να επιβεβαιώσουμε πως εγώ φυσικά δεν εκπροσωπώ όλες τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Εγώ ανήκω στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ που ε, ε, έχει αρμοδιότητα για τέσσερις από τους πέντε οργανισμούς υπό απαλλαγή σήμερα. Ωστόσο παρακολουθώ προσεκτικά τη διαδικασία απαλλαγή, αλλά και σε επίπεδο συμμετοχής μας στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Παρακολουθούμε την καλή εκτέλεση των προπολογισμών, όλες τις πτυχές που ουσιαστικά είναι σημαντικές σε θέματα χρηστής διαχείρισης. Και θα ήθελα να επιμείνω, γιατί για τη δική μου γενική διεύθυνση ΣΑΝΚΟ είναι πολύ σημαντικό. Παρακολουθούμε διαρκώς αδιάκοπα της προόδου των οργανισμών όσον αφορά τις δηλώσεις ε, διένεξης συμφερόντων και συμφερόντων γενικότερα. Έχουν σημειωθεί σημαντικέ πρόοδοι, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Επίσης είναι ένα θέμα όπου πρέπει να αφοσιώνονται διαρκώς οι οργανισμοί. Εμείς επιβλέπουμε τις πρόοδους αυτές των οργανισμών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο για τους οργανισμού όσο και για εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεση, κατάθεση τροπολογιών 19 Δεκεμβρίου 10 η ώρα στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος 24 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού 18 Μαρτίου θα γίνει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση και περνάμε τώρα στο τελευταίο σημερινό σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η Συμφωνία Ναγκόγια Κουαλουμπούρ για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το συμπληρωματικό πρωτόκολλο για Συμφωνία Ναγκόγια Κουαλαλούμπου σε σχέση με την ευθύνη για την αποζημίωση του πρωτοκόλλου Καρθαγένης για την βιοασφάλεια. Αυτός όλος ο τίτλος Τόσου πολλού συναδέλφου, δηλαδή κανέναν δεν τον κινητοποίησε να καταθέσει ούτε μια τροπολογία, αδιαφόρησαν όλοι. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου και έτσι λοιπόν γνωρίζοντα περί τίνο πρόκειται το πρωτόκολλο της Καρθαγέννη για την βιοασφάλεια για την βιοπικιλότητα είναι μια διεθνή συμφωνία που την προστασία των ε, ζώντων οργανισμών ε, σε σχέση με τις ρυθμίσεις που πρέπει να ισχύουν μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης ρυθμίζονται οι διαφορετικές διατάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση πρέπει να διασφαλιστεί ότι μια χώρα πριν από την αδειοδότηση εισαγωγής τέτοιων ζώντων οργανισμών θα πρέπει επαρκώς να ενημερώνεται και να πληροφορείται και εν πλήρη γνώση των επιπτώσεων των αποφάσεων να λαμβάνει σχετικά, σχετική απόφαση. Στο πρωτόκολλο αναφέρεται η, η ρήτρα της πρόνοιας ή πρόβλεψης όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και πάλι επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη οσον αφορα τα θεματα ασφαλειας και παλι επιβεβαιωνεται αυτη η αρχη της πρόνοιας. Επίσης προβλέπεται ένας τομέας ενημέρωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους οργανισμούς αυτούς, τους ζώντες οργανισμούς και για να βοηθά τις χώρες να υλοποιούν το πρωτόκολλο αυτό, την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Και σε σχέση με την δική μου εμπλοκή να πω ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο Ναγκόγια Κουαλαλούμπουρ για τις ευθύνες ε, και την αποζημίωση συνεισφέρει σημαντικά οι στόχοι τη Συμφωνίας για τη Βιοπικιλότητα και του πρωτοκόλου της ε, Καρθαγένης για την βιοπικιλότητα να μπορούν να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν όπως και η οδηγία για την οικολογική υπευθυνότητα για το περιβάλλον, για την οικολογική ευθύνη. Ασχολείται αυτό το πρωτόκολλο με, ειδικά με ευθύνες και αποζημιώσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Είμαστε υπέρ, είμαι υπέρ της απόφασης του Συμβουλίου που εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσυπέγραψε το πρόσθετο πρωτόκολλο της Ναγκόγια Κουαλαλούμπουρ όσον αφορά τις αρμοδιότητες και την έγκριση από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χαιρετίζω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο και ζητεί να επικυρωθεί αυτή, να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωση το δυνατόν γοργότερα. Αυτά είχα να πω. Τώρα ζητώ να αναφέρουν ποιοι συνάδελφοι θέλουν να παρέμβουν. Άννα Ρόσμπαχ παρακαλώ, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι πρέπει να προσυπογράψουμε αυτό το συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Όμως ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις Όσον αφορά ενδεχόμενες ε, ζημίες, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία έτσι ώστε αυτές οι ζημίες να μην περάσουν τα σύνορα, όπως έλεγες και εσύ προηγουμένως. Πρέπει και εδώ να ε, βλέπουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να τις ανταλλάσσουμε. Και βεβαίως και αυτή η αρχή της ε, πρόνοιας είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως εξίσου σημαντική είναι και η ανάγκη νομοθέτησης ε, ε, ορθής ε, κατά την άποψή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να γίνουν με σωστό τρόπο. Και βεβαίως εδώ δεν μιλάμε μονάχα για τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για χώρε ολόκληρου του κόσμου. Εδώ μιλάμε για τρίτες χώρες. Και επομένως αυτό είναι καινούριο και μας ευχαριστεί. Αυτό ήθελα να σα πω. Σα ευχαριστώ πολύ. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως την Εστονία, την Ελλάδα και τη Μάλτα μπορούμε να τις κινητοποιήσουμε να προσυπογράψουν και αυτές αυτό το πρωτόκολλο η Τσεχική Δημοκρατία, η Λετωνία και η Σουηδία έχουν επικυρώσει αυτό το πρωτόκολλο. Περισσότεροι πρέπει να το κάνουν. Καλό θα ήταν αυτό. Είναι πρωτοπόρο αυτή η κατεύθυνση και έτσι το είδαν οι συνάδελφοι. Γι' αυτό δεν έχουμε τροπολογίε και αύριο θα έχουμε σύντομη περίοδο ψηφοφορία επ' αυτού. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε σήμερα. Φτάσαμε στο τέλο των σημείων τη ημερήσια διάταξη για σημερινή μα ημέρα. Θα συναντηθούμε αύριο στι 10 θα επανέλθετε. Οι συντονιστέ στι 9 αλλά θα είναι και κλεισμένων των θυρών συνεδρία των συντονιστών. Και αύριο θα ξεκινήσουμε αμέσω στι 10 με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ θερμά όλου. Και ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους, για τις συναδέρφους και συναδέρφους που άντεξαν μέχρι το τέλος αυτής της συνεδρίασης. Και σε όλους εύχομαι καλό βράδυ. Καλή βράδυ, αύριο θα τα ξαναπούμε. Γεια.